Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο, την κυρία Βέσταγερ, στην ανταλλαγή απόψεων για τον διαφθορωτικό διάλογο με την ΕΚΟΝ. Είναι ο πρώτος για το 2017 ακολουθεί τις ψηφοφορίες τις οποίες κάναμε το μήνα Φεβρουάριο στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού. Και διεξάγεται η συνάντηση αυτή μια θλιβερή ημέρα θα έλεγα, ένα χρόνο μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που τιμήσαμε σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε και την πρόταση οδηγίας για την ενίσχυση των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών να είναι ισχυρότερες και να διασφαλίσουν την εσωτερική αγορά της, την, να ενισχύσουν την εσωτερική αγορά. Είναι μεικτή αρμοδιότητα. Ξέρετε ότι είχαμε κάνει ένα σεμινάριο γύρω από αυτό το θέμα στα πλαίσια της συναπόφασης έναν τομέα ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος θα έλεγα για τη σωστή λειτουργία της ε, ενιαίας αγοράς. Ευχαριστούμε λοιπόν την Επίτροπο για τις προτάσεις της, την ευχαριστούμε για τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει για να μας κάνει μία πρόταση συναπόφαση στον τομέα του ανταγωνισμού. Θα σας δώσω το λόγο τώρα επίτροπε και μετά θα έχουμε τις ε, κανονικές συζητήσεις μας. Μάργαρετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που είπατε και για την θλιβερή αυτή επέτειο. Ένας χρόνος από τις τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες ε, πραγματικά θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει φυσικά να τιμήσουμε, να αποτίσουμε φόρο τιμή σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν και που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τα φρικτά αυτά γεγονότα. Εμείς σαν Ευρωπαίοι πολίτες, σαν όργανα, σαν κράτη-μέλη, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να διαδηλώνουμε εναντίον της τρομοκρατίας υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας. Σε τρεις μέρες καλούμεθα να εορτάσουμε τα 60 χρόνια της συνθήκης της Ρώμης. Αυτό είναι κάτι που έθεσε τα θεμέλια για μια εξαιρετική μορφή συνεργασίας, όπως επίσης και για την ενιαία αγορά γνωρίζετε και θα συμφωνήσετε μαζί μου λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε τον ανταγωνισμό για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές στην Ένωση. Να διασφαλίσουμε στους καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα σε ανεκτές τιμές. Αλλά φυσικά αυτό δεν είναι μόνο δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίθετα από το 2004 μέχρι το 2014 το 85% των αποφάσεων για τον ανταγωνισμό έχουν ληφθεί όχι από εμά αλλά από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ε, είναι σημαντικό οι αρχές αυτές να είναι ισχυρές έτσι ώστε να μπορούν οι χώρες να υποφελούνται από διαδικασίες οι οποίες είναι δημιουργές απασχόλησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν οι αρχές αυτές να έχουν όλες τις εξουσίες τις οποίες χρειάζονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια γιατί θεωρούμε πράγματι ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτή τη διπλή νομική βάση, να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί το εκλογικό σώμα των κρατών μελών έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές επί του ανταγωνισμού αρχές έχουν τα μέσα τα οποία απαιτούνται έτσι ώστε να εφαρμόσουν και να επιβάλλουν τους κανόνες και τους νόμους για τον ανταγωνισμό και να μην μπορεί κανείς να διαφύγει στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Αν τυχόν δραστηριοποιείται σε μία χώρα μπορεί να ανοιχνεύεται και να επιβάλλονται οι κυρώσεις που είχαν προβλεφθεί και στην προηγούμενη. Ζητήσατε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις τέτοιες έτσι ώστε οι εθνικές αρχές να έχουν τις απαιτούμενες εξουσίες. Όπως είπα τώρα πια έχουμε την πρόταση εδώ. Πήγαμε αρκετά γρήγορα θα έλεγα. Βέβαια χρειάστηκε κάποιος χρόνος γιατί ε, προϋπήρξε, μεσολάβησε, διαβούλευση με το κοινό ε, και από την ήρθαν επαφές και από ε, οργανώσεις καταναλωτών και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι τα προγράμματα αυτά επί τα οποία οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο να λειτουργούν σωστά έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τι μεταχείριση θα τύχουν, αν ας πούμε αναφέρουν ένα καρτέλ. Η πρόταση διασφαλίζει οι αρχές αυτές να έχουν το προσωπικό και τα χρήματα για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κάτι το οποίο τους δίδει και τις απαιτούμενες νομικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας για να μην επηρεάζονται από τους πολιτικούς, από τις κυβερνήσεις αλλά να κάνουν τη δουλειά τους, οι οποίες, ε, να κάνουν δουλειά τους με σωστό τρόπο. Πρέπει επίσης να απομακρύνουμε και τα εμπόδια τα οποία παρεμποδίζουν τις εθνικές ευχές ε, από το να καθορίζουν πρόστιμα, έτσι ώστε να το σκέφτονται δύο φορές οι επιχειρήσεις αν παραβιάζουν τον νόμο. Φυσικά όταν έχει κανείς αυξημένες εξουσίες αποκτά και αυξημένες ευθύνες Όλες οι αρχές του προϋπολογισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους με σωστό τρόπο, σεβόμενοι και τα δικαιώματα υπεράσπισης των επιχειρήσεων. Συνεπώς λοιπόν, μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας, με το τέλος μάλλον αυτής της διαδικασίας, οι καταναλωτές στο σύνολο της Ευρώπης θα μπορέσουν να ωφεληθούν πλήρως από τον ανταγωνισμό για να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά και όταν λέω να λειτουργήσει σωστά, δεν αναφέρομαι μόνο σε καλές τιμές και σε επιλογή, αλλά για σε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Μια άλλη, ένα άλλο θέμα από την έκθεση, το οποίο μας απασχόλησε πρόσφατα, είναι το πόσο ο ανταγωνισμός θα βοηθήσει και τους γεωργούς. Οι κανόνες δεν κρατούν μόνο τις τιμές χαμηλές για τους καταναλωτές υπερασπίζονται τον ανταγωνισμό και στις αγορές από τις οποίες εξαρτώνται οι γεωργοί. Ε, νωρίς φέτος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση της Επιτροπής ε, για το καρτέλ ε, στους, σε συγκεκριμένες συνθετικές ζωοτροφές και υπήρξε ένα πρόστιμο 175 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, στην περίπτωση των φωσφορικών ζωοτροφών. Ε, επίσης εξετάζουμε και τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων έτσι ώστε οι καταναλωτές να μην βγαίνουν χαμένοι από αυτές. Και πολλές φορές οι πελάτες αυτοί είναι οι γεωργοί. Θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα οδηγήσουν οι συγχωνεύσεις σε αύξηση των τιμών και δεν θα αποτρέψουν επιχειρήσεις να εργαστούν για νέα προϊόντα τα οποία να είναι ασφαλέστερα για τους γεωργούς και το περιβάλλον. Φυσικά το μέλλον των Ευρωπαίων γεωργών δεν είναι μόνο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν έτσι ώστε οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις να είναι πιο κερδοφόρες όταν σαν παράδειγμα συνδυάζονται. Ε, συνεργαζόμενοι σε οργανώσεις παραγωγών μπορούν να επεξεργάζονται, να αποθηκεύουν και να διανέμουν μαζί τα προϊόντα τους. Έτσι μπορούν να γλιτώσουν χρήματα, να προσθέσουν αξία και αυτό είναι κάτι που θα αυξήσει γενικότερα τα έσοδά τους. Αν το κάνουν αυτό σε αρκετά ευρύ ε, πλαίσιο, θα γίνουν οι επιχειρήσεις τους πιο ανθεκτικές και θα μείνουν χαμηλά οι τιμές για τους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και ένα χρόνο ε, κυκλοφορήσαμε κατευθυντήριες γραμμές ε, για γεωργούς που παράγουν ε, ελαιόλαδο, βοηδή και αρρώσιμα προϊόντα έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Μαζί με τον Επίτροφο Χόγκαν προσπαθούμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε οι κανόνες του ανταγωνισμού να είναι πιο απλοί και καλοί για τους γεωργούς. Να μου επιτρέψετε να πω τώρα λίγα λόγια για τις κρατικές επιδοτήσεις. Εμείς προσπαθούμε εδώ και χρόνια να επεξεργαστούμε τις απαιτήσεις έγκρισης. Θέλουμε να διευρύνουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε General Block Exemption Regulation, τον κανονισμό δηλαδή γενικών εξαιρέσεων, όπως επίσης και τον πίνακα αποτελεσμάτων για, όταν βλέπουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές επιδοτήσεις βλέπουμε ότι έχουμε κάνει βήματα πρόοδου. Το 2013 το 1 τρίτο των νέων μέτρων κρατικής βοήθειας είχε χρειαστεί την έγκρισή μας εκ των προτέρων. Αυτά το 2013. Τώρα ο αριθμός αυτός έχει πέσει στο 4% που απαιτείται έγκριση πριν εφαρμοστεί. Με τη διεύρυνση για μια ακόμη φορά του κανονισμού λοιπόν και καλύπτοντας λιμένες και μικρούς αερολιμένες θα μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το ποσοστό έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να προωθούν τις ιδέες τους ε, το ταχύτερο δυνατόν και ε, όταν δίδονται κρατικές επιδοτήσεις να δίδονται με αποτελεσματικό τρόπο. Δουλεύουμε επίσης ε, για να δούμε πού το δημόσιο χρήμα δεν θεωρείται κρατική βοήθεια. Το προηγούμενο καλοκαίρι δημοσιεύσαμε ε, ένα επεξηγηματικό σημείωμα για την έννοια της κρατικής επιδότησης ή βοήθειας. Το σημείωμα αυτό εξηγεί το τι μετράει σαν βοήθεια και κυρίως αυτό που δεν μετράει σαν βοήθεια και δεν απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, πήραμε μία σειρά αποφάσεων τα τελευταία δύο χρόνια να, για να δείξουμε πότε οι τοπικές ε, υποδομές θεωρούνται κρατική επιδότηση γιατί δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Σαν παράδειγμα ένας μικρός Ολλανδικός λιμίν ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τοπικούς αλληλείς γαρίδας ή ε, ένα μικρό λιμανάκι στο, στο, στην ίσο Φερ στη Γερμανία για τον πληθυσμό 8.000 κατοίκων. Έχουμε όμως και άλλες περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται ο κίνδυνος από τις υποδομές αυτές τρέβλωσης του ανταγωνισμού. Για τα υπόλοιπα όμως δεν έχουμε να κάνουμε με κρατικές επιδοτήσεις. Λοιπόν, προσπαθούμε να βγαίνουμε από τη μέση, από τη σκηνή, όταν δεν απειλείται σοβαρά ο ανταγωνισμός και μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη εκεί όπου χρειάζεται και το κάνουμε αυτό ε, για να είμαστε ταχείς και αποτελεσματικοί. Όπως είπα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε περιπτώσεις ε, οι οποίες ε, βοηθούν, σαν παράδειγμα υποστήριξη με συγκεκριμένα ευεργετικά φορολογικά μέτρα οι χώρες μέλη αποφασίζουν το πώς θα δαπανίσουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Η δουλειά μας είναι αυτό να μην βλάπτει τον ανταγωνισμό. <coughs> Φυσικά για να ελέγχει την κυβέρνηση το κοινό χρειάζεται ενημέρωση. Και γι' αυτό είναι οι κανόνες μας για την διαφάνεια σημαίνουν ότι κάθε ε, κρατική βοήθεια άνω των 500.000 ευρώ θα πρέπει να δημοσιεύεται online δείχνοντας το ποιος πήρε πόσα. Τους 9 μήνες που πέρασαν 1.700 τέτοιες περιπτώσεις έχουν δημοσιευθεί και όλοι είναι, ε, έχουν την δυνατότητα να δουν ακριβώς τι έχει γίνει. Αυτό ε, επίσης σημαίνει ότι κάθε κρατική βοήθεια ανάνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ κατέτος θα πρέπει να αξιολογείται για να βλέπουμε αν πράγματι πετυχαίνει τους στόχους της. Τα κράτη-μέλη στην φάση αυτή εξετάζουν και αξιολογούν 33 προγράμματα, αξία συνολικά 38 δίσκα κατέτος. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές να κάνουν ε, την σωστή δουλειά στην προστασία της του ανταγωνισμού. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και από κοινού και μεμονωμένα κάνουμε εταιρικέ σχέσεις έτσι ώστε η κρατική βοήθεια που δίδουν να μην υπονομεύει τον ανταγωνισμό. Και όπως είπα, αυτό είναι και ο λόγος και η βάση θα έλεγα των προτάσεων που έχουμε υιοθετήσει σήμερα, έτσι ώστε οι εθνικές αρχές να έχουν πραγματικές εξουσίες στα χέρια τους. Είναι μια ιδέα που αυτή η Επιτροπή έχει υποστηρίξει με σοβαρό τρόπο. Χαίρομαι λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο προωθώντας τις ιδέες αυτές και είμαι στη διάθεσή σας για να εξετάσουμε μαζί τις λεπτομέρειες. Και φυσικά περιμένω και να ακούσω τις απόψεις σας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Ήδη χθε κατανείμαμε τις αρμοδιότητες ε, για τον εισηγητή και την ομάδα της διαπραγμάτευσης. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία για να έχουμε και το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ας ξεκινήσουμε με τον ε, Μάρκους Φέρμπερ, που είναι όχι μόνο ε, Πρόεδρο τη Επιτροπή αλλά και τη Ομάδα Εργασία για τον Ανταγωνισμό. Μάρκο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την πρόταση την οποία υποβάλλατε σήμερα και στην Ομάδα Εργασία μα θα ασχοληθούμε και στην Επιτροπή θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία ε, κάνετε και έχουν σχέση με τι Εθνικέ Επιτροπέ Ανταγωνισμού, γιατί αυτό προσδίδει ποιότητα στι εργασίε μα και χαιρετίζουμε αυτή την ε, πρωτοβουλία. Έχω Τρία σχόλια. Πρώτον, Μαδέρα, Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την Πορτογαλική Αυτόνομη Περιοχή της Μαδέρα έχει επιτρέψει ένα, πολύ, ένα καθεστώς φορολογικό με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Κάναμε σχετική έρευνα για το θέμα και είδαμε ότι η Μαδέρα λειτουργεί λίγο σαν τις Μπαχάμες και τον Παναμά. Το 2020 θα πρέπει να γίνει επανεξέταση, αναθεώρηση αυτού του καθεστώτος. Τι έχετε να σχολιάσετε για αυτές τις έρευνες, λοιπόν. Δεύτερον, η διεθνής διάσταση του δικαίου ανταγωνισμού. Η Επιτροπή με τον Καναδά έχει συνάψει μία συμφωνία παρόμοια με αυτή που έχουμε με την Ελβετία και μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε σχετικές ε, πληροφορίες γιατί δεν έχει επικυρωθεί αυτή η συμφωνία και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να επικυρωθεί από τον Καναδά. Και τρίτο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια έχει λάβει κάποιες αντιφατικές αποφάσεις όσον αφορά την ασφάλεια των καταθέσεων και τον ανταγωνισμό. Αυτό έχει σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να γίνει με τα μέσα των καταθετών. ποια είναι τα μέτρα και οι κανονισμοί για την προληπτική εποπτεία. Ε, το Φεβρουάριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την ετήσια έκθεση για την Τραπεζική Ένωση ανέφερε προς την Επιτροπή ότι θα πρέπει να εξετάσει τους κανόνες για τις ε, εθνικές ενισχύσεις σχετικά με ένα σύστημα εγγύσεων και προληπτικών μέτρων. Νομίζετε ότι η Επιτροπή θα ανταποκριθεί σε αυτή την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Uh, on the first question of... Για την πρώτη ερώτηση για τη Μαδέρα. Η ιδέα του να έχουμε μία ελεύθερη ζώνη ε, αποσκοπεί στο να βελτιώσουμε την ανάπτυξη της ε, περιφέρειας αυτής. Βέβαια πρέπει να τηρούμε τους κανόνες των ε, κρατικών ενισχύσεων και με τις πληροφορίες που προκύπτουν ε, παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε σε επαφή με τις πορτογαλικές αρχές για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Του του λεχθέντος, ίσως να πρόκειται για μη κρατικέ ενισχύσεις και να πρόκειται απλώ για φοροδιαφυγή, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες φορολογικέ αρχές. Δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει γιατί ακόμη διερευνούμε το θέμα. Για το δεύτερο θέμα, για την ε, Συμφωνία Συνεργασίας Δευτέρας Γενεάς με τον Καναδά, χαίρομαι διότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και το επόμενο βήμα θα είναι να δώσει την έγκριση στο Συμβούλιο και να υπογράψει τη Συμφωνία και στη συνέχεια θα σταλεί στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που βρίσκεται θετική αυτή την συμφωνία και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο πιέζει ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν για το τρίτο θέμα, για τις τράπεζες και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων έχουν ως πρόθεση να είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μέχρι 100.000. Δεν έχουμε μεγάλη πρακτική εμπειρία για να δούμε τι γίνεται αν υπάρχει ένας καθαρά ιδιωτικός μηχανισμός. Δεν είναι σε αυτή την περίπτωση δικό μας θέμα να αποφασίσουμε πώς γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων, αλλά θα πρέπει να είναι ιδιωτικός αυτός ο μηχανισμός. Αν είναι κατόπιν κρατικής διάταξης ή αν εμπλέκεται το κράτος, τότε μπαίνουμε στις κρατικές ενισχύσεις. Δεν είναι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο το θέμα αυτό του συστήματος εγγύησης καταθέσεων και δεν ξέρω αν υπάρχει τελευταία ενημέρωση την οποία δεν έχω. Έχω περισσότερο χρόνο, λέει ο κύριος Φέρμπερ. Δυστυχώς όχι. Δεν είχαμε βάλει το ρολόι εξ αρχής και αν φαίνεται ότι έχετε χρόνο είναι γιατί δεν έχει ρυθμίσει το ρολόι. Κύριε Μπεχές. Ε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε στην υπόθεση της Apple η Ιρλανδική κυβέρνηση ε, ε, έκανε καταγγελία για την ε, απόφαση αυτή και 14 σημεία θεώρησε ότι δεν στέκουν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε την εντύπωση ότι η μάχη θα είναι μεγάλη και ίσως θα μπορούσατε να Ενημερώσετε το κοινοβούλιο μας που βρισκόμαστε ακριβώς και ποια προβλέπετε ότι θα είναι στο μέλλον η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τα θέματα των ε, α, αλγόριθμων και των, α, ε, της τεχνητής νοημοσύνης Google την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο εκφράσατε την ανησυχία σας για το θέμα αυτό και διαπιστώνουμε ότι στη ΣΥΠΑ, στο αντίστοιχο κλάδο, εξελίσσεται μια αντίστοιχη τεχνολογία και θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε πώς εκτιμάτε στο μέλλον τη δράση σας. Για να μην υπάρχει τεχνητή διαμόρφωση των τιμών για τη χρήση τέτοιων αλγορίθμων ε, τεχνητής νοημοσύνης της ε, Google. Μου φαίνεται ότι πρόκειται ε, βασικά για θέμα πόρων. Μήπως όμως πίσω από αυτό κρύβεται και θέματα πρακτικών, προβληματικών πρακτικών, τις οποίες ε, θα μπορούσατε ήδη να αντιφρυνήσετε στο Κοινοβούλιο. Όπως είπατε και η Apple και η Ιρλανδική κυβέρνηση έκαναν καταγγελία για την δικαστική αυτή απόφαση. Το χρονοδιάγραμμα Τη υπόθεση προφανώς θα καθοριστεί από το δικαστήριο. Δεν ξέρω κατά πόσον θα πάρει πολύ ή όχι. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί για να υπερασπίσουμε τη θέση μας με τον πιο δυναμικό τρόπο που γίνεται. Για προφανείς λόγους. Ενδεχομένω να υπάρχει και λιγότερο κίνδυνο ε, καταγγελίας, γιατί κάθε τέτοια υπόθεση έχει αντιστοιχεί ποιότητα και σημασία στην ομολογία, μια και πρόκειται για μια ένωση που βασίζεται στο κράτο δικαίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό προφανώ. Συνεργαζόμαστε με του Ιρλανδού σε ό,τι αφορά την ανάκτηση, γιατί πρόκειται για μεγάλα ποσά. Η ανάκτηση για τη Fiat και τη Starbucks έχει ήδη γίνει και έχει γίνει η καταγγελία και έφεση. Τώρα τα πράγματα είναι τα ποσά αυτά σε κλειστούς λογαριασμούς, έχει γίνει η ανάκτηση. Είμαστε λοιπόν, θεωρώ, σε καλό σημείο σε ό,τι αφορά τις εταιρείε ε, του συστήματος, οι οποίες θα πρέπει να ξανακοιτάξουν τους φόρους τους για κάθε μία ξεχωριστά. Αλλά το κάνουν και νομίζω ότι πηγαίνει καλά η διαδικασία τώρα. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Apple, φυσικά συνεργαζόμαστε με την Ιρλανδία για να το πετύχουμε αυτό, είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η ανάκτηση του τουλεχθέντος. Προφανώς θα πρέπει να δούμε πώς θα τα κρατήσουν τα χρήματα αυτά, γιατί προφανώς ενδεχομένω να πάρει πάρα πολύ χρόνο μέχρι ότου αποφασιστεί η τύχη των χρημάτων αυτών. Για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις όταν ε, παραγγέλνουν ή καταρτίζουν ε, αλγοριθμούς να έχουν υπόψη τους και θέματα σηματότητας. Είναι, μου προκαλεί πάντα έμπνευση το γεγονός ότι ακούω ανθρώπους που δουλεύουν στον τομέα της ιδιωτικής σφαίρας να ξέρουμε ότι η ιδιωτική σφαίρα δεν είναι κάτι το οποίο προστίθεται στο τέλος, καπάκι. Όχι, είναι κάτι το οποίο διατρέχει όλη την δουλειά και θα πρέπει να έχει ξεκινήσει από την αρχή. Το ίδιο ισχύει και για του αλγορίθμου. Και προφανώ όσο πιο πολλά ποσά έχουμε, τόσο πιο σημαντική και ε, σημαντική θα είναι η αλγορίθμη αυτή. Γιατί τελικά το αποτέλεσμα θα το νιώσει ο κόσμο. Ω τώρα δεν έχουμε δει ακόμα αλγοριθμού που να συνεργάζονται ή να βρουν ανεξάρτητα για καθορισμό τιμών. Αυτό είναι πάντα ανθρώπινου, ανθρωπογενές, ανθρώπινης προέλευσης. Επίσης, αν τίθεται θέμα τεχνητής νοημοσύνης που έχει καθορίσει τιμές, πάντα θα ευθύνεται τελικά κάποιος, ε, κάποια επιχειρήση, κάποια εταιρεία, κάποιο άτομο. Ως τώρα δεν έχουν γίνει σχετικές έρευνες. Αλλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Και καλά κάνουμε και το διευκρινίζουμε. Σχόλια εκτό μικροφώνου. Ναι, έχει ξεκινήσει η συζήτηση στη ΣΥΠΑ και θα έπρεπε να ξεκινήσει και εδώ, στην Ευρώπη, η συζήτηση να αντιληφθούμε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των εργαλείων IT. Πώς θα τα προστατεύσουμε κιόλα και πώς θα εγγυηθούμε το θέμα της συμβατότητας, τι θα γίνει με τις ανησυχίες των πολιτών και ασφαλώς έχει ξεκινήσει η συζήτηση πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση για να μην χάσουν τελικά οι πελάτες. Ευχαριστώ. Λέρνερ. κομισάρι. Ευχαριστώ. Την ευχαριστώ λοιπόν για τον αγώνα που δίνει για, τον ανταγων... για την προφύλαξη του ανταγωνισμού από ε, παράνομες φορολογικές καταστάσεις. Είναι αξιολόγο το ότι μπορούμε εμείς να ε, θεωρούμε τις αδικαιολόγητες φοροαπαλλαγές σαν απαράδεκτες ε, κρατικές επιδοτήσεις. και βλέπουμε το τι ακριβώς έχει γίνει σε χώρες όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, με μεγάλες επιχειρήσεις στα πλαίσια των επιθετικών τους φορολογικών πολιτικών. Έχει σημασία λοιπόν πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά για το σύνολο της Ένωσης και καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε και ποιο θα είναι το μελλοντικό καθεστώς. να μας πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας για τα αποδεκτά επίπεδα φορολογίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα για την Apple και την Starbucks βλέπουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν προταθεί. Αυτές θα είναι οι τελευταίες παρεμβάσεις σας ή θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες. Να σας ρωτήσω επίσης αν έχετε όλη την απαραίτητη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για τις έρευνες που κάνατε για αυτές τις συγκεκριμένες προσπάθειες. Υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια. Σας ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά σας λόγια, για τη δουλειά που κάναμε μέχρι τώρα, το εκτιμώ δεόντως. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή. Το μέσο για την κρατική βοήθεια είναι κάτι το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή σου όπου παρουσιάζονται επιλεκτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και όπου ε, έχουν τεθεί σε αμφισβήτηση πόροι που προορίζονται ε, για το κράτος. Φορολογικές ευνοϊκές ρυθμίσεις, προφανούς μερικές φορές ε, χαρακτήρα που μπορεί να χαρακτηριστούν κρατική βοήθεια. Έχει υπάρξει καθοδήγηση τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να παραμείνουν εκτός της παράνομης επιδότησης και προσπαθούμε να δώσουμε όσο περισσότερη κατεύθυνση μπορούμε, όσο αυξάνεται η εμπειρία μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ βλαβερό οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τη φορολογία τους, τους φόρους τους και να βλέπουν κάποιες άλλες που δεν πληρώνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο φύγει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της επιχειρήσεις όταν βλέπουν ότι άλλοι δουλεύουν και στην ουσία εν μέρη πληρώνονται από τα χρήματα των φορολογουμένων. Εδώ θα έλεγα είναι ένας τομέας στον οποίο και με τις προσπάθειες του Πιέρ Μοσκοβισή μπορούμε να προχωρήσουμε. Να υπάρξει σαν παράδειγμα μια κοινή επιχειρηματική βάση επιβολής. Σε δύο-τρεις χώρες στην αρχή τουλάχιστον για να δούμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει και θα είναι πιο δύσκολο για τις μεγάλες επιχειρήσεις να αποφεύγουν να πληρώνουν φόρους. Νομίζω επίσης ότι η διαφάνεια είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε σαν πολίτες να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει με τις επιχειρήσεις, εάν πράγματι συνεισφέρουν, όπως και πράγματι κάνουν οι περισσότερες, στην κοινή προσπάθεια στις κοινωνίες μας. Νομίζω ότι ο σκελετός της οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πληρώνουν φόρους, προσλαμβάνουν σταζιέρ, μαθητευόμενους μάλλον και γι' αυτό θα πρέπει εάν παράνομες μορφές επιδότησης δίδονται, να βρούμε ποιες είναι και να επιβάλλουμε κυρώσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω, λέει ο κύριος Τρεμόζα ή Μπαλσέλς. Θα αναφερθώ στην περίπτωση της βάρος της Google και θα σας ρωτήσω πράγματα τα οποία σας είχα ζητήσει και την εποχή που παρουσιαστήκατε εδώ τον Οκτώβριο του 2014. Εδώ και 7 χρόνια είπε η Επιτροπή ότι μπορεί να υπάρχουν θέματα αντιτράστ με την Google. Είπατε επίσης ότι ε, θα υπάρξει έλεγχος και για την Κάσμπρομ, με την οποία όμως κλείσατε τη διαδικασία μετά από κάποια χρόνια. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο και με την Google. Μιλάτε επίσης για το δικαίωμα υπεράσπισης των δικηγόρων της Google. Φυσικά, σε 7 χρόνια το δικαίωμα υπεράσπισης δεν είναι κάτι το οποίο έγινε αρκετά σεβαστό. Και τέλος οι υπηρεσίες σας ε, ε, ολοκλήρωσαν τα στοιχεία που σας έδωσε η Google. Όπως γνωρίζετε ε, υπάρχουν άλλες εταιρείες όπως το Yelp και τα λοιπά που αναγκάστηκαν να κλείσουν διότι ήταν τέτοια η συμπεριφορά της Google. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια φαινόμενα δημιουργούν μονοπόλια και γι' αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να πάρετε ε, μέτρα, αποφάσεις και ίσως ε, και τον επόμενο μήνα να μας ανακοινώσετε κάτι τέτοιο εδώ. Τέλος, δεν γνωρίζετε να γνωρίζουμε τους μυστικούς αλγόριθμους της Google ή τη σύνθεση τη μυστική της Coca-Cola. Θέλουμε όμως κάποια στοιχεία από τις υπηρεσίες της Google. Έχει το 92% της αγοράς και η αγορά αυτή αυξάνεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι τελικά όποιος επικρατήσει στην αρχή επικρατεί συνεχώς. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να ανακοινώσω κάτι στην επόμενη συνάντηση και στο Σικάγο, διότι δεν θα πάω στο Σικάγο, αναγκάστηκα να ακυρώσω. Όχι εξαιτία σας πάντως. Για την Google συγκεκριμένα, Έχουν γίνει πάρα πολλές ε, συζητήσεις για εξωτερικού τύπου ρυθμίσεις και αν ο Αλμούνια ήταν επιτυχής, τότε δεν θα υπέφεραν πάρα πολλές ε, επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους διαδικασίες υπήρξαν αλλά απέτυχαν. Θα ήταν πραγματικά πετυχημένο το να πετύχαιναν οι διαδικασίες αυτές, γιατί επαναλαμβάνω ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν θα υπέφεραν όπως υπέφεραν. Εμείς επεξεργαζόμαστε τις απαντήσεις της Google στις ερωτήσεις μας, στη δήλωση αντίρρησης που κατέθεσε η Google, Και όπως γνωρίζω δεν ξέρω αν η υπόθεση αυτή θα πάει στη δικαιοσύνη ή όχι, αλλά οποιοδήποτε που έχει μια υπόθεση να ρυθμίσει με την Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει την ποιότητα της διαδικασίας και το δικαίωμα υπεράσπισης που έχει, γιατί αλλιώς αυτό θα υπονόμευε την δουλειά την οποία κάνουμε. Συνειδητοποιώ επίσης το ότι Έχουμε να κάνουμε με, ε, παγκόσμιες, ε, με παγκόσμια φαινόμενα διεθνών επιχειρήσεων. Ε, δεν είναι μόνο η Google βέβαια, είναι και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι η Google παραμένει κυρίαρχη ακόμα και όταν η χρήση του διαδικτύου γίνεται από κινητά και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη στιγμή ανάλογα με τις ε, αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν χρησιμοποιούμε ε, κινητά μέσα να ε, γνωρίζουμε ποιος παρέχει την υπηρεσία. Κοιτάξτε, η Επιτροπή έχει δυνατότητες και αρμοδιότητες να παρέμβει, να το κάνετε γρήγορα. Ε, θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας. Λόπες Βεμέιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Επίτροπε για τη διαθεσιμότητά σας για μια ακόμη φορά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα βασικά. Καταρχάς τις αγροτικές αγορές και την αγορά του ηλεκτρισμού μετά από τις ανακοινώσεις που κάνατε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας σήμερα, αυτά που είπατε για τη Γεωργία. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα μας δώσατε και τις απαντήσεις σας στην προηγούμενη έκθεση για τον ανταγωνισμό. Αναφερθήκατε στην δεσμευτική δράση για τις καταχρήσεις στην τροφιμική αλυσίδα. Έχουμε να κάνουμε με μια βιομηχανία πολύ συγκεντρωτική σε επίπεδο input και σε επίπεδο ολιγοπολίων όπως τα ζυζανιοκτώνα και ταυτόχρονα με την περίπτωση της Μονσάντο και στην περίπτωση της εμπορίας, κάτι το οποίο φύγει διπλά τους καλλιεργητές. Θα πρέπει λοιπόν η αρχή ανταγωνισμού να τα συζητήσει αυτά και στο τέλος του 2016 δημιουργήθηκε, κυκλοφόρησε μια έκθεση γύρω από τις καταχρήσεις των τομέα των τροφίμων. Ε, ποια είναι η κατάληξη αυτών των συζητήσεων και τι θα κάνετε για να προστατεύσετε τους μικρούς παραγωγούς και τους γεωργούς στον τομέα του ηλεκτρισμού για να ολοκληρώσω και τη δεύτερη ερώτησή μου, σε μια γραπτή ερώτηση που καταφέσαμε ε, ζητάμε εξηγήσει ε, για την απότιμη αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιανουάριο στην Ισπανία, στο Βέλγιο και στη Γαλλία δυστυχώς πολλές φορές τις γραπτές ερωτήσεις αποφεύγει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς πιστεύουμε ότι η φιλελευθεροποίηση των αγορών του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί σε καταστάσεις εναντίον της βάρος του ανταγωνισμού, που είναι δύσκολο να τις εντομετωπίσει κανείς και δεν μπορεί να διακρίνει τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις εθνικές αγορές και στο σύνολο των ενοποιημένων αγορών. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να αυξήσουμε την παρουσία των δημοσίων αρχών, όπως επίσης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εθνικοποίηση των ολιγοπολίων, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους τους οποίους οι ρυθμιστικές αρχές δεν κατάφεραν να λύσουν, όπως ο καθορισμός των βιομηχανικών τιμολογίων και η ενεργειακή φτώχεια. Δύο διαφορετικές ε, παρατηρήσεις όσον αφορά τους γεωργούς. Είπα και στην αρχή ότι προσπαθούμε να δώσουμε ως το δυνατόν πιο συγκεκριμένα στοιχεία, καθοδηγώντας τους αγρότες για το πώς μπορούν να ε, ενώσουν τις προσπάθειές τους για θέματα αποθήκευσης και βελτίωσης της συλλογικής τους παραγωγικότητας, για να έχουν ε, μεγαλύτερη επίπτωση στην αλυσίδα αξίας. Εξετάζουμε θέματα συγχωνεύσεων που μπορεί να δημιουργούν ακόμη περισσότερο τα θέματα εισρώων και γι' αυτό είναι σημαντικό για τους πελάτες μας, τους αγρότες στη συγκεκριμένη περίπτωση, να υποφελούνται του ανταγωνισμού, όχι μόνο ε, σε θέματα τιμών και ποιότητας, αλλά και σε θέματα καινοτομίας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για την καινοτομία να υπάρχουν ουσίες που δεν είναι επικίνδυνες είτε για τους ίδιους τους αγρότες είτε για το περιβάλλον. Υπάρχει λοιπόν συγκέντρωση στα θέματα εισρώων, πάρα πολλοί αγρότες και συγκέντρωση και πάλι στη λιανική πώληση και κάποια ενδιάμεσα στάδια μέχρι τους ε, καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να φτάσουν αυτοί οι κανόνες μέχρι τους αγρότες, να τους αναγνωρίζουν και να τους χρησιμοποιούν. Γιατί ένας αγρότης χρειάζεται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα φτιάξει κάτι και πώς θα το κάνει να λειτουργήσει. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να προσλάβει δικηγόρους για να τον βοηθήσουν ή ακόμη και αν προσλαμβάνουν οι αγρότες δικηγόρους και εκείνοι δεν ξέρουν εύκολα πώς θα δράσουν. Αλλά εμείς θέλουμε να δώσουμε οδηγίες, σαφέστερες οδηγίες και συγκεκριμένες οδηγίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα οποία προσφέρονται. Δεύτερον, πριν από λίγους μήνες, όπως είπατε, είχαμε μια έκθεση και τώρα με τον Φιλ Χόγκαν, τον Επίτροπο Υπεύθυνο για Θέματα Γεωργίας, προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. ο ανταγωνισμός είναι κάτι καλό, αλλά θα πρέπει να είναι και λειτουργικός, να, να ωφελεί και εμάς τους ίδιους, όχι να ωφελείται μόνο η αλυσίδα ε, αξίας, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αναβλήθηκε μια συνάντηση, αλλά θα επανέλθουμε και το παρακολουθούμε. Για, τον, ε, για την ηλεκτρική ενέργεια, οι ρυθμιστές πρέπει να ρυθμίσουν τα στοιχεία της αγοράς για να αποφύγουν να θέμει το ανταγωνισμό. Υπάρχουν ιδέες για την απελευθέρωση της αγοράς, αλλά θα πρέπει να είναι απελευθερωμένη, να είναι ρυθμισμένη η αγορά για να μπορούν να υποφεληθούν οι πελάτες. Οι γαλλικές αρχές προσπάθησαν ε, να επιβάλλουν ένα πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ στην ε, ε, εταιρεία NG νομίζω, αλλά δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα σε άλλες αγορές, στη δική σας αγορά παραδείγματος χάρη. Μια αρχή ανταγωνισμού θα πρέπει να φροντίσει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών όταν υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές. Η Ενεργειακή Ένωση έχει ως έννοια το ότι δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στην εθνική αγορά γιατί η ηλεκτρική ενέργεια ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα και μπορούμε να υποφεληθούμε και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειάζονται βέβαια επενδύσεις και θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε και τα θέματα μεγάλων εχμών ε, κατανάλωσης, για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα θέματα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με ε, τρόπο ε, εφικτό. Μιχαήλ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την Επίτροπο. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, τον έλεγχο των συγχωνεύσεων. Όταν η Facebook εξαγόρασε την WhatsApp, δεν εξετάστηκε αυτή η εξαγορά, γιατί δεν υπήρχαν πολλοί στη WhatsApp, υπήρχε μια βάση πελατών, αλλά δεν υπήρχε αγορά. Αυτό ίσως δεν ισχύει για την ψηφιακή αγορά. Οι κανόνες είναι σχεδόν απειρχαιωμένοι. Εδώ και 12 χρόνια έχουμε κανόνες για την ψηφιακή αγορά. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέους κανόνες και θα προωθήσετε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, Ε, θέματα ταχύτητας. Δουλεύετε αρκετά γρήγορα και εσείς και οι υπηρεσίες σας. Αλλά εγώ είμαι ανυπόμονο. Με το που ξεκινάτε κάτι, περιμένω αμέσω αποτελέσματα. Και ιδίω στην ψηφιακή οικονομία, πάντοτε είναι πήγοντα τα θέματα. Νομίζετε ότι οι τρέχοντε κανόνε σε επιτέχουν να έχετε την επιθυμητή ταχύτητα ή θα έπρεπε να επιταχύνουμε τι διαδικασίε. Ιδίω όταν μιλάμε για τον κανονισμό, ε, για τη συνεργασία με, εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ. ρυθμιστικές αρχές. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται κάποια προσαρμογή. Τρίτον, για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Βλέπω ότι σιγά σιγά οι 28 κυβερνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιε από αυτέ τουλάχιστον ε, επανέρχονται σε εθνικές εγωιστικές πολιτικές δίνοντα πλεονεκτήματα σε εθνικές εταιρείε. Εγώ βλέπω μια αυξητική τάση του τελευταίους μήνες και φαντάζομαι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί. Ποιο είναι ο ρόλο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και ποιο θα είναι στο μέλλον. και πώς ε, μπορούμε να έχουμε κάποια εγγύηση ότι δεν θα καταληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοιου είδους εγωισμούς. Σας ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτηση, για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή εξέτασε ε, την συγχώνευση Facebook και WhatsApp, διότι μας ε, παρεπέμφθη το θέμα από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να δούμε το θέμα και ήδη στην πρώτη φάση ε, συμμετέσχομεν. Είχαμε κάνει μια ένσταση είχαμε την ανησυχία ότι δεν μας έδωσαν επαρκή πληροφόρηση για τη συγχώνευση για να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία σχετικά με τους χρήστες και τη συγχώνευση στοιχείων των δύο οντοτήτων. Τώρα μας έχει απαντήσει η Facebook ε, στην κοινοποίηση των δικών μας αιτιάσεων και για μας έχει κέρια σημασία το να έχουμε σαφή πληροφόρηση. Γιατί αν δεν έχουμε σωστή πληροφόρηση δεν μπορούμε να καταβάλουμε την προσπάθεια που θα θέλαμε. Μπορεί να μην αλλάζει το αποτέλεσμα της συγχώνευσης, αλλά θα έχουμε τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για το πώς μπορούμε να έχουμε τις σωστές συγχωνεύσεις με ορατό τρόπο, κάναμε δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους, γιατί ίσως να μην έχουμε το επαρκές κατόφλι για να μπορούμε να εξετάσουμε μία συγχώνευση. Μπορεί δηλαδή μια εταιρεία να έχει πληροφόρηση, γνώση και στοιχεία τα οποία είναι κάτω από το κατόφλι αλλά πολύ σύντομα θα φτάσουν σε ένα πολύ ψηλότερο κύκλο εργασιών και τότε θα είναι ώρα τι για μας αυτή η συγχώνευση. Εξετάζουμε τις απαντήσεις που πήραμε από τη διαβούλευση για να δούμε αν μπορούμε να εκπονήσουμε κανόνες. Γιατί οι κανόνες μας προσπαθούμε να είναι όσο δυνατόν περισσότερο αντικειμενικοί και όχι τυχαίοι για να δουν ε, οι εταιρείε ε, αν συμφωνούν με αυτά τα οποία προτείνουμε. Και για την ε, τελευταία σα ερώτηση, δύο ερωτήσεις μάλλον είχατε. μία ερώτηση ήταν για την ταχύτητα. Όντω οι κανόνε μας επιτρέπουν να λειτουργούμε αποτελεσματικά, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τμήματα της διαδικασίας, γιατί ακόμη και αν κερδίσουμε μια εβδομάδα σε κάποια σημεία θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας ταχύτερα. Και κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε ε, και στην πρόταση για τους NTAs είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε μια πολύ αυστηρή προσέγγιση στην Επιτροπή, δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεται ε, αμετάκλητη ζημία που είναι πολύ δύσκολο και σπάνιο να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σε κάποιες νομολογίες στην Γαλλία χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και επιτυχημένα. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας, αφήνοντας και το δικαίωμα υπεράσπισης και ταυτόχρονα αν μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε ασφαλιστικά μέτρα. Και τελευταία σας ερώτηση για, τις, για την νομική εγγύηση είναι κάτι που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Είχε προκύψει και παλαιότερο όταν ο προκάτοχός μου εξέταζε τη δομή εξουσίας μετά από 10 χρόνια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού για να έχουμε τις νομικές εγγύησεις ότι μπορούμε να έχουμε ε, ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και θα αντικατοπτρίζονται όλες οι πτυχές της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ, Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ τον, την Επίτροπο που είναι ανάμεσά μας σήμερα. Μία ερώτηση τι διαβεβαιώσεις μπορείτε να μας δώσετε για τους ε, καταθέτες οι οποίοι έπεσαν θύματα απάτης στην Ιταλία και αν θα υπάρξουν ε, αποζημιώσεις σε περίπτωση bail-in και burden sharing. Δεύτερη ερώτηση, κάπως πιο περίπλοκη. Το 2008 μέχρι το 2013 πολλές χώρες χρησιμοποίησαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να βοηθήσουν τις τράπεζές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αναζητήσει να δει τι στρεβλώσεις δημιουργούνται με βάση ε, τις ε, παρεμβάσεις που έγιναν υπέρ των τραπεζών τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα επίσης οι δημοσιογράφοι οι Ιταλοί αναφέρθηκαν σε αυτούς που χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα στις ε, τράπεζες. Αυτό δεν οφείλεται σε μικρούς δανειολήπτες, αλλά στους λεγόμενους ε, ε, μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, δανειολήπτες που μπορεί να είναι βιομηχανικές εταιρείες κτλ. και εκπρόσωποι της πολιτικής. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αξιολογήσει τι συνέπειες κοινωνικές είχαν σε πάρα πολλές χώρες οι βοήθειες που δόθηκαν σε τράπεζες από το 2008 μέχρι το 2013 και όταν έχει αμφιβολίες να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να κάνουν ελέγχους γιατί από ό,τι φαίνεται οι πρακτικές αυτές δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχείς Υπάρχει μια συνέργεια ανάμεσα σε μεγάλους επιχειρηματικούς κύκλους, πολιτικούς και ε, ηθήνοντες τραπεζών. Uh, Για την πρώτη ερώτηση των ασφαλείων για τους μικρούς αποταμιευτές. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό, γιατί προφανώς αν έχει κάποιος αποταμιεύσεις ε, στην τράπεζα και ακούει διάφορες φήμες, ε, θέλει να ενημερωθεί. Όσο υπάρχει αποταμίευση, είναι πάρα πολύ καλό, θεωρώ, το ότι υπάρχει ο κανόνας ότι καλύπτεται κανείς για τις πρώτες 100.000, ότι υπάρχει εγγύηση. Το θέμα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μ, κάποια παρανόηση, γιατί νόμιζε κανείς ότι κάνει αποταμίευση και ότι έχει έναν λογαριασμό αποταμίευσης, αλλά στην ουσία έχει ένα τμήμα της τράπεζας και μετά ότι της έκπληξη αποκαλύπτεται ότι αν θέλει να... Ότι υπάρχει η έκθεση αυτή και του λένε, για παράδειγμα, στους πελάτες ότι αν θέλει να ωφεληθεί από τα πλέον θα πρέπει να διακινδυνεύσει και λίγο. Και υπάρχει λοιπόν μια τέτοια προώθηση λανθασμένων πρακτικών για τις πωλήσει. Και τα κοιτάμε αυτά σε ό,τι αφορά τις δικασίες κυρίως ε, των κρατικών επιδοτήσεων προκειμένου να μην χρειαστεί να αποζημιωθούν άτομα τα οποία θα έπρεπε να είναι ενήμερα για το γεγονός ότι αναλαμβάνουν ρίσκο αλλά η καταπολέμηση τέτοιων ε, λανθασμένων πρακτικών πώληση θεωρώ ότι είναι σημαντική. Και στο Κοινοβούλιο έχετε περάσει νομοθεσία η οποία ουσιαστικά ο σκοπό έχει να διευκρινίσει το τι έκθεση έχει ο πελάτη στην τράπεζα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, αρρωγή προς τις τράπεζες, τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφήρμοσε τότε την νομοθεσία. Όταν ένα κράτος μέλος βρέθηκε σε μια κατάσταση και χρειάστηκε να ληφθεί η δράση για την τράπεζα. 122 περιπτώσεις έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τραπεζών που βρίσκονται σε φάση εξυγίανσης ή τακτικής ε, απομείωσης. Και αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της ε, κρατικής, των κρατικών επιδοτήσεων, για παράδειγμα. Τέλος, για το ερώτημα που θέσατε για τα ονόματα. Αυτό δεν το εξετάζουμε. Εμείς εξετάζουμε το πώς μπορεί να συσταθούν τα προγράμματα, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία. Ήταν, μεγάλη εταιρεία, ήταν μια μεγάλη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ήταν ενεργή στον τομέα των ακινήτων. Και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό για τα επόμενα χρόνια. Και εκεί που τα πράγματα περιπλέκονται σε ό,τι αφορά τα δάνεια αυτά, τα οποία δεν αποδιδουν no non-performing loans, είναι όταν γίνεται αυτό σε διάφορου τομεί. Γιατί τα δάνεια αυτά στο παρελθόν ήταν κυρίω στη, στα κινητά. Τότε θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μια εταιρεία διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα κατέχει το θέμα. Αν υπάρχουν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όμως τέτοια δάνεια που δεν αποδίδουν, δεν είναι είναι προφανές ότι θα υπάρχει μία μόνο εταιρεία διαχείρισης πλησιακών στοιχείων. Και αυτό θεωρώ ότι αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο τα τελευταία χρόνια και προφανώς το αντιλαμβανόμαστε. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα κρατήσει κάποια κράτη-μέλη τα δάνεια αυτά που δεν αποδίδουν. Αποτελούν και ένα βαρύδι στην οικονομία. Και γι' αυτό λοιπόν συστήνονται τέτοιοι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν τα δάνεια αυτά. Με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να καταστούν ένα εργαλείο χρήσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χόκμαρκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας και για την προβολή που δώσατε στην πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνάδει πολύ με το ότι, ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις ξεχνάμε τι ακριβώς ε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει, τι σημαίνει για την καθημερινή οικονομική μας ζωή. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Για το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την νομική βεβαιότητα, καταρχάς σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα. Νομίζω ό,τι και να λέμε για τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για την κρατική επιδοτήσεις, για τις φορολογικές, ε, τα φορολογικά συστήματα. Το πρόβλημα είναι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιβάλλει πρόστιμα αναδρομικά για 10-20 χρόνια πριν σε εταιρείε. Πείτε μας λοιπόν η αναδρομικότητα. Τι σημαίνει αυτό και για την νομική βεβαιότητα για τους επενδυτές και για την προσαρμογή τους στους κανόνες των μεμονωμένων χωρών. Κατά δεύτερον, κάτι άλλο. Η ανάγκη είναι να αναδειχθούν κάποιοι Ευρωπαίοι πρωταθλητές σε παγκόσμιο προσκήνιο. Μπορεί να είναι άδικο αυτό που λέω, αλλά υπάρχει μια τάση. Οι παγκόσμιοι ηγέτες από μικρές χώρες να την χάνουν διαφορετική αξιολόγηση από ότι οι παγκόσμιες ε, ηγετικές εταιρείε από μεγάλες χώρες που κάνουν συγχωνεύσεις. Παρά το γεγονός ότι όλοι δρούν στην ευρωπαϊκή και στην τοπική τους αγορά. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό σήμερα, σε ό,τι αφορά το μέλλον δηλαδή. Και μια τελευταία ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχτεί τις ρυθμίσεις αυτές που αναφέραμε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το Nord Stream 2. Είναι σημαντικό λοιπόν το να μιλήσουμε και για αυτά που έχουμε ήδη πετύχει, όχι μόνο για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι βασικό στην πολιτική. Μιλάμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε στο μέλλον, ξέρετε συχνά. Αλλά θεωρούμε δεδομένα αυτά που έχουμε ήδη πετύχει. Εδώ λοιπόν στην 60η επέτειο της Συνθήκη της Ρώμης θα ήθελα να πω το γεγονό ότι και μόνο το γεγονό ότι έχουμε 70 χρόνια ειρήνη ε, δεν είναι επειδή δεν υπάρχουν πλέον καθόλου πόλεμοι και ότι δεν υπήρχε καμία, κανένα έναυσμα για πόλεμο. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα συνέβαινε αυτό. Και ας μην το παίρνουμε ως δεδομένο. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Ας το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο. Αυτό ας μας δώσει την έμπνευση, τη δέσμευση που χρειάζεται να λύσουμε τα σημερινά προβλήματα. Η νομική βεβαιότητα προκύπτει όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ένα στόχο με διαφορετικού τρόπου. Κυρίω με μία απόφαση ως επιτοπλίστων. Δεν ε, υπήρξε, για παράδειγμα, κοινοποίηση των συστημάτων σε ό,τι αφορά ε, τη φορολόγηση των ε, επιχειρήσεων. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει εγκριθεί, αλλά αν θέλει κανεί να υποβάλλει τα συστήματα αυτά προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε μόνο υπάρχει απόλυτη νομική βεβαιότητα. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόζει το εθνικό, την εθνική νομοθεσία που αποφασίζεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτά τα δύο θα πρέπει να συμβαδίζουν. Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη αναδρομικότητα σε ό,τι αφορά την ανάκτηση κρατικών επιδοτήσεων. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι έχουν αλλάξει εκ των υστέρων οι κανόνε και αυτό είστε όλοι βουλευτέ. Είναι, ξέρετε, η εξαίρεση. Όταν γίνεται αυτό, μάλιστα, γίνεται για να ωφελήσει κάποιον. Εδώ μιλάμε για φόρου που δεν έχουν καταβληθεί. Δεν είναι πρόστιμα. Είναι φόροι που δεν έχουν πληρωθεί. Και 10 χρόνια πίσω μπορούμε να πάμε από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να ερευνούμε το θέμα. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί σωστό και δέοντα τρόπο αντιμετώπιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά του παγκόσμιου πρωταθλητέ τη εταιρεία αυτέ στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κανένα κανόνα να μην είναι μεγάλη μια εταιρεία. Μπορεί να μεγαλώσει όσο θέλει, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει το μέγεθό τη. Και τι εξετάζουμε όταν εξετάζουμε περιπτώσει συγχωνεύσεων, γιατί έχουν γίνει μεγάλε συγχωνεύσει και πρόσφατα. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο πελάτη μπορεί να στραφεί κάπου αλλού. Αν η κοινή, ο κοινό όμιλο αυξήσει τι τιμέ, μπορεί ο καταναλωτή να πει εντάξει λοιπόν, εγώ παίρνω το καπλάκι μου και πάω αλλού. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει ακόμα ανταγωνισμό. Σε κάποιε περιπτώσει όμω δεν βγάζει νόημα. Σε ό,τι αφορά τι τηλεπικοινωνίε, για παράδειγμα, αν ε, αυξηθούν οι τιμέ στη χώρα σου, τι θα κάνει, θα γραφτεί σε διπλανή χώρα. Ακόμα και με τις αλλαγές που έγιναν με την υπεριαγωγή. Και όλο και πιο πολλές αγορές κατίστανται ευρωπαϊκές και παγκόσμιες. Αυτό προφανώς δημιουργεί με ένα μεγάλο περιθώριο για ευρωπαϊκές εταιρείε για το Nord Stream 2. Ξέρετε ότι ο συνάδελφος Σεύκοβιτς και Κανιέτα είναι οι αρμόδιοι και είναι στη φάση ακόμα που εξετάζουν το κατά πόσο διαφορετικές νομικές βάσεις ε, εφαρμόζονται και ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση. Ελπίζω να καταλήξουν συντόμως σε κάποιο συμπέρασμα, ωστόσο. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Τσάνι. And I pass the chair to Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη διαθεσιμότητά σας, ακόμη και όταν συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις μας επάπειρον. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στις 25 Μαρτίου δεν είναι ότι μόνο υπεγράφει η συνθήκη της Ρώμης, αλλά και η συνθήκη Ευρατόμ. Και η συνθήκη αυτή ρυθμίζει ακόμη τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ατομική ενέργειας, παρότι πιστεύω ότι πριν από 60 χρόνια οι ανανεώσιμες ενέργειες ε, δεν ήταν γνωστή έννοια. Η συνθήκη Ευρωτόμ ορίζει ότι αν ένα κράτος μέλος, όπως το δικό μου, η Ουγγαρία, θέλει να ε, δημιουργήσει ένα πυρηνικό σταθμό, θα στραφεί στην Επιτροπή για να τη βοηθήσει να βρει την πλέον κατάλληλη μέθοδο. Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει το πράσινο φως στην Ουγγρική κυβέρνηση να δημιουργήσει το νέο πυρηνικό σταθμό στην Ουγγαρία που παρελθόντος είναι ρωσικής τεχνολογίας του περασμένου αιώνα, αναστάτωσε πάρα πολύ και ανησύχησε πάρα πολύ τον πληθυσμό της Ουγγαρίας. Η πλειοψηφία των πολιτών στην Ουγγαρία δεν θέλουν την πυρηνική ενέργεια. Η κυβέρνηση συνεχίζει όμως να έχει την ίδια πρόθεση. Ξέρω ότι μόνο οι Ούγγροι μπορούν να αλλάξουν την κυβέρνηση, ελπίζω κάποια μέρα, αλλά οι σημερινές αποφάσεις ε, θα έχουν και πλέον μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δεν κατηγορώ ούτε εσά ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατανοώ τους κανόνες. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι ικανοποιημένος από την αποφασή σας. Θέλω να σας υπενθυμίσω μία πτυχή του θέματος που ίσως δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη. η Ουγγρική κυβέρνηση απαγορεύει σαφώς σε ορισμένους ανταγωνιστές τη συμμετοχή στην αγορά. Δεν εκδίδουν πλέον άδειες ε, για ε, έργα αιωλικής ενέργειας και επιβάλλουν ε, αυστηρούς φόρους στις ε, ανανεώσιμες ενέργειες για να ετοιμάσουν το δρόμο για την πυρηνική ενέργεια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν ε, είναι χαμένη υπόθεση ή αν έχετε την πρόθεση να παρακολουθήσετε το θέμα. Η κυρία Φερσάγκερ. Όπως είπατε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τους κανόνες και έχετε παρακολουθήσει αυτή την προθεση να παρακολουθησετε το θεμα κυρια φερσαγκερ από κοντά. Για μένα είναι κάπως δύσκολο, διότι προσωπικά δεν είμαι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Δεν έχουμε στη χώρα μου και καλά κάνουμε. Βέβαια το ενεργειακό μείγμα είναι επιλογή του κάθε κράτους μέλους και της κυβέρνησης του κάθε κράτους μέλους και αυτό το σέβομαι. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορούν το αν μπορεί η κυβέρνηση να λάβει μια απόφαση αλλά για το αν υπήρξε εθνική ενίσχυση, κρατική ενίσχυση. Σε τέτοια περίπτωση ένα κράτο μέλο, η Ουγγαρία σε συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να αναλάβει δεσμεύσει για να μην πλήττεται ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν κάνει. Η συνάδελφος Εξβιέτα Βιανκόφσκα εξετάζει τι διαδικασίε δημοπράτηση για να δει εάν όντως στηρίθηκαν σωστέ διαδικασίες. Και ο συνάδελφος ε, Κανιέτε εξετάζει το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας. Αν ε, οι ε, ρυθμιστικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα να εξετάσουν και θέματα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Ουγγρικής κυβέρνησης. Για αυτά που αναφέρατε για την μία έκδοση αδειών για αιωλική ενέργεια, για νέες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας ή για επιβολή φορολογίας στις ανανεώσιμες ενέργειες, εάν υπάρξει μία καταγγελία, την εξετάζουμε. Όχι μόνο για θέματα εθνικής ε, κρατικών ενισχύσεων, αλλά εάν παρεμβαίνει η για επιβολη φορολογιας στι ανανεωσιμε ενεργειες εαν υπαρξει μια καταγγελια την εξεταζουμε οχι μονο για θεματα εθνικης κρατικων ενισχυσεων αλλα εαν παρεμβαινει η κυβερνηση στην αγορά, βεβαίως και πρέπει να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. αλλά Μασού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για την εξαιρετική σας παρουσίαση και συγχαρητήρια ε, για τι δράσει σας. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση ε, όσον αφορά το πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, χωρίς ε, καμία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς προσωπικά, κάθε άλλο. Αναφέρατε στην εισαγωγική σας παρουσίαση τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Μία ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής Ανταγωνισμού είναι το διοικητικό της καθεστώς. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται, αλλά είναι ανεξάρτητη από πολιτικές ε, εξουσίες από, με επιρροές από την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Από την εμπειρία έχουμε δει ότι ε, είναι λαμπρές οι δράσεις της, ιδίως με μια λαμπρή επίτροπο όπως είστε εσείς. Παράλληλα όμως ε, μπαίνουμε σε μια λεπτή κατάσταση, διότι θα μπορούσαν να σας κατηγορήσουν ότι εξυπηρετείτε ε, ένα είδος βιομηχανικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να σας κατηγορήσει κανείς ότι δεν υποστηρίζετε επαρκώς την οικονομική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας είστε μέλος, αλλά ως αρχή ανταγωνισμού είστε και ανεξάρτητοι. Πιο μακροπρόθεσμα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι θα απαιτεί το μία αλλαγή των συνθήκων για κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού δεν θα μπορούσε στο μέλλον να είναι πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μην ε, υπόκειται σε τέτοια δίκη προθέσεων και να θεωρείται όπως η Αμερικανική Αρχή FTC. Well, Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία θα πρέπει να συζητηθεί επαρκώς και συχνά. Οι ανεξάρτητες αποφάσεις στην ουσία είναι θα έλεγα αυτό το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους θα επιβληθεί ο σεβασμός του ανταγωνισμού. Ισχύει απόλυτα στην περίπτωσή μου. Αν δεν το τηρήσω αυτό νομίζω ότι θα θέσω σε αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε την επιβολή του νόμου. Μέχρι τώρα από πλευρά του ECDA δεν έχει υπάρξει η αδίποτε αναφορά σε πιθανή έλλειψη αντικειμενικότητας. Τηρούμε και ελέγχουμε και θέματα όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πράγματα ως προς αυτό έχουν όπως θα έπρεπε να είναι. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην σύνταξη της πρότασης την οποία έχετε πλέον μπροστά σας Προσπαθούμε να σεβαστούμε πλήρως ε, την διοικητική αν θέλετε ιστορία και κουλτούρα κάθε χώρας και ταυτόχρονα προσπαθούμε να προτείνουμε να υπάρχουν ισχυρότερες αρμοδιότητες και ισχυρότερες εφαρμοστικές δυνατότητες γιατί όπως είπατε εργάζονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο οι ελεγκτικές αρχές επί του ε, ανταγωνισμού σε κάθε χώρα. Και αυτό ισχύει και για τη δική σας χώρα. Έχουν ανεξαρτησία, έχουν ανεξάρτητο τρόπο σκέψης και ελευθερία να δουλέψουν όπως θα έπρεπε να ε, το κάνουν και το κάνουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα προωθείται ακόμα περισσότερο μέσω των νομικών εγγυήσεων τις οποίες εμείς επιζητούμε. Δέχομαι όμως ότι υπάρχει μια πρόκληση. Η πρόκληση αυτή είναι να είμαστε πάντα πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον φάκελο του ανταγωνισμού τονίζοντας όμως ότι μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί ε, σε αμφισβήτηση η αντικειμενικότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Νίνα έχει το λόγο. Um, τώρα για τις αρχές της εθνικής επί του προϋπολογισμού. Πράγματι θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες των αρχών αυτών και η ανεξαρτησία του FDA είναι κάτι το κομβικό. Τι μηχανισμό θα έχετε στη διάθεσή σας έτσι ώστε να υπάρξει συμβατότητα ανάμεσα στις αποφάσεις που λαμβάνονται στον τομέα της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού. Δεύτερη ερώτηση. Βασική προτεραιότητα είναι η επένδυση σε αγορές high-tech υψηλής τεχνολογίας. Είναι εγγύηση αυτό, με, συμφωνώ με αυτό. Διάβασα όμως ότι η Ρωσική Αρχή επί του προϋπολογισμού αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Apple ε, συμφώνησε με άλλες επιχειρήσεις ε, για να κρατήσουν υψηλά τις τιμές των φορητών τηλεφώνων, των κινητών συγγνώμη τηλεφώνων. Ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι έχουν περιθώρια κέρδους τεράστια σε κάθε ε, συσκευή την οποία πολλούν οι της Apple. Ένα άλλο θέμα Ξέρετε η Χάινεκεν η οποία είναι ε, πολυεθνική θέλει να εξαγοράσει μία από τις παλιότερες αγγλικές εταιρείες pub στις, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε επίσης ότι έτσι θα αποκτήσουν πρόσβαση στην κατανάλωση ζήθου. Ξέρετε ότι ο ζήθος είναι σημαντικότατο στη χώρα μου. Τίθεται θέμα ανταγωνισμού προς αυτό σε πολλές χώρες είναι σημαντική η κατανάλωση του συγκεκριμένου ποτού. Για πάρα πολλά χρόνια όταν πήγαινε κανείς στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης είχαν ένα τεράστιο, μια τεράστια αφίσα με τον μπουκάλι τους που έλεγε σας καλωσορίζουμε στην πιο χαρούμενη χώρα στον κόσμο. Τώρα είμαστε η δεύτερη χαρούμενη αλλά πού θα πάει θα πάρουμε τη θέση των Ορβηγών όπου να είναι. Τώρα για την συγχώνευση αυτή που είπατε δεν τη γνωρίζω. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, θα το ελέγξουμε αλλά δεν ξέρω να σας πω πότε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές είναι το ότι ανήκουμε στο ίδιο δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού είναι θα έλεγα ένα δίκτυο χαμηλό σε επίπεδο διοικητικών πρωτοκόλων και υψηλό σε επίπεδο παραγόμενης ουσίας. Α, περιπτωσιολογικά εξετάζουμε θέματα και συγκεκριμένους τομείς έτσι ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα χαρακτήριζα πολύ σημαντικό. Φυσικά έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες αλλά οι ευθύνες αυτές ε, θα έλεγα ε, αποδίδονται με δίκαιο τρόπο, με διαφανή τρόπο και λόγω και της αναγνώρισης της προσπάθειας η οποία έχει γίνει από τις εθνικές αρχές. Αν δεν το έκαναν αυτό οι εθνικές αρχές δεν θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν θα προστατεύαμε τους πολίτες όπως θα έπρεπε. Έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης έτσι ώστε αν μια εθνική αρχή ασχοληθεί με μια υπόθεση ε, που έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον οι αποφάσεις ε, για το ποιος θα ασχοληθεί με την υπόθεση να λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν αν θα είναι δηλαδή ευρωπαϊκού επίπεδου η αντιμετώπιση του προβλήματος ή εθνικού επίπεδου. Το πιο σημαντικό τώρα <clears throat> σε σχέση με την επίπτωση στις τιμές των προϊόντων είναι ότι υπάρχουν πραγματικά διαφορές ε, στις διάφορες χώρες και πράγματι θα ήταν καλό να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες χρήσης ε, επιχειρήσεων και τύπων προϊόντων από ό,τι έχουμε σήμερα σε ορισμένες χώρες, σαν παράδειγμα η Apple, είναι πάρα πολύ ψηλά. Ε, σε άλλες χώρες ε, το σύστημα λειτουργικό Android είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, οπότε η Apple δεν είναι σημαντική. Ιβάνα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την Επίτροπο σας Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σα και τι καλές απαντήσει. Η ε, δική μου ερώτηση έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση της Κροατίας και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις αθνιστικές αρχές συνταγωνισμού, σε ό,τι αφορά ε, τις εξαγορές ε, ε, στη βιομηχανία. Πρόκειται για μικρές εξαγορέ, μικρού όγκου, χωρί μεγάλο αντικτύπο, στη Νότιο Δαλματία, μία περιοχή η οποία είναι συγκρίσιμη σε μέγεθος και έκταση με την Ιντανέζικη περιοχή της Νόρτιλα και έχουμε κύκλο εργασιών 4, εκατομμύρια ευρώ. Μικρός κύκλος εργασιών. Φυσικά, σκόπος της αρχής ανταγωνισμού μας είναι να εξασφαλίσει την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Καλύτερες τιμές, πιο, πολύ, ε, πιο πολλές επιλογές για τους πελάτες, αλλά και πιο πολλή ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, όπως είπατε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση η Κροατική Αρχή Ανταγωνισμού που παρακολουθούσε την υπόθεση εδώ και καιρό είναι αντίθεστη με την αξιολόγηση της Digicomt σε ό,τι αφορά θέματα ουσίας και νομολογίας και θεωρεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και ότι θα πρέπει να επιτραπεί αυτή η εξαγορά. Πρόκειται για ένα καινούριο κράτο μέλο, όπου έχουμε την αίσθηση ότι καταρακώνεται η εμπιστοσύνη στου ευρωπαϊκού θεσμού. Αυτή η λειτουργία είναι προβληματική, λες και αγνοούν μεν τους δε. Ελπίζω η λύση να μην βρεθεί στα δικαστήρια, γιατί η αρνητική απόφαση στην παρούσα φάση ουσιαστικά θα αναβάλει την, ε, τις επενδύσεις στην Κροατία, την επένδυση στην Κροατία και την εξαγορά και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλη την αγορά, σε όλη την ε, οικονομία. Η Επιτροπός. Να πω ότι, κοιτάξτε, είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση, συγκεκριμένη και δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Η νομική προθεσμία νομίζω εκπνέει στις 18 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε ε, αρμοδιότητα για την ε, υπόθεση αυτή. Όντως αφορά την Δαλματία μόνο, αλλά αφορά μία πολύ μεγάλη τσιμεντοβιομηχανία. Με μεγάλο ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Στη Δαλματία λοιπόν επικεντρώνεται η εταιρεία αυτή, αλλά είναι μεγάλες εταιρείε αυτές. Δεν είχε υπάρξει κάποια καταγγελία τότε όταν ε, αποφασίσαμε να εξετάσουμε την υπόθεση. Αργότερα εκφράστηκαν αμφιβολίες από την εταιρεία κατά πόσον είχαμε αρμοδιότητα ή όχι. Οι κροατικές ε, αρχές δεν έκαναν αυτά που έπρεπε τότε και γι' αυτό λοιπόν στράφηκαν σε μας. Και λυπάμαι που λέτε ότι δεν σας ακούμε, γιατί μπορεί να μην συμφωνούμε στην εκτίμηση και στην αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά θεωρώ ότι είναι καλή η επικοινωνία. Και προφανώς ακούμε καλά και μας ακούν, ελπίζω, και οι κρατικές αρχές. Είναι σημαντικό να υπάρχει input και από τις αρχές. Και προφανώς η διαφωνία για την αρμοδιότητα ίσως να είναι πιο σημαντική και από την ίδια την υπόθεση στην ουσία της. είναι σημαντικό γιατί αφορά το τσιμέντο και είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση σε κανονικές τιμές γιατί το τσιμέντο έχει ιδιαίτερο ρόλο στην τοπική βιομηχανία και από ό,τι ξέρετε το τσιμέντο δεν μπορεί να ταξιδέψει και να μεταφερθεί και ιδιαίτερα μακριά. Είναι μάλλον τοπικό προϊόν. Τέλος. Είχαμε διάφορες υποθέσεις που αφορούσαν το τσιμέντο τα τελευταία χρόνια και προφανώς εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα και στην προκειμένη περίπτωση όπως και σε άλλες συγχωνεύσεις Και πάντα σκοπός ήταν να υπάρχει ακόμα ανταγωνισμό ε, στην αγορά και να υπάρχουν και επιλογές και τιμέ λογικές. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες δικασίες σε όλη την Ευρώπη. Είτε πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι της Ευρώπης, είτε για μεγάλα κομμάτια της Ευρώπης. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Φέρπερ, ο Αλφρέντ ε, τελευταίο. Τρει ερωτήσει, πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Για δεύτερη διαθεσική χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ετήσια έκθεση της για τον ανταγωνισμό ζήτησε διαχωρισμό αυστηρό των ε, υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταρτίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και αυτών που ευθύνονται για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών. Έχετε οποιοδήποτε σχέδιο προγραμματίζετε να αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτή την έλλειψη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ανταγωνισμού, σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτούς που θέτουν, εφαρμόζουν και ελέγχουν τις αρμοδιότητες αυτές. Κατά δεύτερον, στην, όταν ε, ακούσαμε την ακρόασή σας εδώ στο Κοινοβούλιο, ως Επιτροπός, είπατε ότι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει τον ανταγωνισμό εξαρτάται από την ικανότητά τη να συνεργάζεται με άλλου φορείς, όπως παραδοσιακούς εμπορικούς φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αναδυόμενες οικονομίες. Πείτε μα λοιπόν, δώστε μα λίγο feedback. Τι πρόοδο έχει σημειωθεί στην πολιτική ανταγωνισμού από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά συμφωνίε και συνεργασίε με τρίτε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο. Στι 9 Νοεμβρίου πέρσι συναντηθήκαμε εδώ στην Επιτροπή για να συναντήσουμε τη συμφωνία με τον Καναδά. Η πρόταση συμφωνίας προέκυψε μετά από 8 χρόνια διαπραγματεύσεων με τις Καναδικές Αρχές. Το 2008 ξεκίνησαν. Οι διαπραγματεύσει αυτέ τώρα δεδομένη τη συμφωνία ΣΥΤΑ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν πιστεύετε ότι η προτεραιότητα είναι να τελειώνει και αυτή η συμφωνία των συντομότερων δυνατών. Um, ναι, όντως ε, ισχύει το ότι άλλα τμήματα ασχολούν με την ε, θέσπιση των κανόνων και άλλα με την υλοποίηση των κανόνων. Κάποια τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης ασχολούνται με τη διαμόρφωση των κανόνων. Υπάρχει ένα τέτοιο εσωτερικό τμήμα. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όταν αλλάζουμε τους κανόνες που χρησιμοποιούμε, παραδείγματος χάρη τον, πρόσφατα για τον κανονισμό των γενικών εξαιρέσεων, κάνουμε διαβουλεύσεις. Είχαμε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για τις ε, γενικές εξαιρέσεις λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία έχουμε αποκομίσει από τους ε, φορείς, ε, τους εμπλεκομένους στα κράτη-μέλη και κάνουμε και μια δεύτερη δημόσια διαβούλευση για να έχουμε την αντίδραση μετά τη δική μας αντίδραση στην πρώτη διαβούλευση. Όταν ε, θεσπίζουμε κανόνες δεν πρέπει να το κάνουμε απομονωμένοι αλλά σε αλληλεπίδραση με την ε, κοινωνία που μας περιβάλλει. Για την ε, παγκόσμια συνεργασία Ξεκινάμε τώρα συμφωνίες δεύτερης γενεάς. Καταρχήν έχουμε συμφωνήσει με τους ομολόγους ε, στην Ιαπωνία να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και σε συγκεκριμένα θέματα προσπαθούμε να έχουμε στενή συνεργασία τέλη Απριλίου θα πάω στην Κίνα και θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Πέρυσι, μετά όμως την ημερομηνία που αναφέρατε, Ετοιμάσαμε ένα έγγραφο σχετικά με τις συγχωνεύσει, για την προετοιμασία των συγχωνεύσεων, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις που κάνουν συγχωνεύσει και για τις κινεζικέ αρχές που ελέγχουν τις συγχωνεύσει, να γνωρίζουν τις διαδικασίες, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής διαφάνεια με τι εμπλεκόμενε επιχειρήσει. Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα για μας να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση κατά προτίμηση εντό του Διεθνούς Δικτύου συνεργασία, ε, όπου διεθνώς δυστυχώς δεν είναι μέλο η Κίνα. Και στα μέσα Μαΐου θα πάω στο Πόρτο για την ετήσια διάσκεψη του δικτύου ανταγωνισμού. Σύμφωνο μαζί σας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε συμφωνία στο Συμβούλιο για να περάσει η Συμφωνία Συνεργασίας Δευτέρας Γενιάς με τον Καναδά και ελπίζουμε με τη δική σας βοήθεια να περάσει και από το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν, διότι έχει σημασία να συνεργαζόμαστε στενά, καθώς με την παγκοσμιοποίηση και με την ταχύτητα που ισχύει στο επιχειρήν, χρειαζόμαστε και εμείς ταχείες διαδικασίες για να μπορούν και οι αρχές ανταγωνισμού να έχουν μία ταχεία αντίδραση σε θέματα ανταγωνισμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ, για την υπομονή σας και για όλες σας ε, τις ε, απαντήσεις. Ήταν μια πληρέστατη ε, συζήτηση ελπίζω να συνεχίσουμε αυτές τις τακτικές επισκέψεις και την καλή μας συνεργασία. Δεν έχουμε χρόνο για, το, για ερωτήσεις κάτω στη Ελπίζω να μην εξήγησα τη δική σα υπομονή, λέει η Επίτροπο. Μερικέ φορέ μακρηγορώ με τι απαντήσει μου και σα ζητώ συγγνώμη. Αλλά οποτεδήποτε με καλέσετε, ευχαρίστω θα έρθω για μια τέτοια ευρία ανταλλαγή απόψεων και πιο συγκεκριμένα για προτινόμενε ε, ε, νομικέ διατάξει σας υπόσχομαι ότι θα αποτελείτε προτεραιότητα για μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε που σύμφωνα με τη μέση διάταξη Περνάμε στην ψηφοφορία και ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Τα ψάχνει να βρει την κάρτα της. Την έχει πολύ ωραία και εγώ έχω τη δική μου. Αλλιώς πώς να προεδρεύσω. Να ελέγξουμε λοιπόν. Ξεκινάμε με έλεγχο των καρτών για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η δοκιμή. Voted. Ivana has not yet voted. Kay has not yet voted. Εψήφισαν όλοι. Προσπαθώ με το ραντάρ μου να πιάσω όσους δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Ωραία. Ξεκινάμε με την πληροφορία για τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματο για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση τη συμμετοχή των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακή πολιτική στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020. Η συγκητή ήταν ο Φίλιπ Λάμπερτ, που δεν είναι σήμερα παρόν. συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Νομίζω ότι γνωρίζετε το θέμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι η... Α, ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Close. τη της ψηφοφορίας. 44 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στην ομάδα που έκανε τις διαπραγματεύσεις. Μετά έχουμε την έκθεση για τη θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020. Θείοντος Στόλογιαν, τον εισηγητή. θέλετε το λόγο. Δεν είστε υποχρεωμένος. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή και ευχαριστώ και τον πρόεδρο, τον κύριο Γκουαλτιέρη, που διεξήγαγε τις διαπραγματεύσει πάρα πολύ σωστά. Ψηφίζουμε λοιπόν και πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Τέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 41 υπέρ, 2 κατά 4 εποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Η επόμενη έκθεση είναι ένα σχέδιο έκθεση για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείε Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητας. Η συγκήτρια η κυρία Σύρβα Πιέτη Κάινεν. Αρχίζουμε με την συμβιβαστική τροπολογία Α. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 131 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά. Υπερβόνς υπέρ, ναι, αποχές. Με χτύπησε η υπερβάνσα, ναι. Φαντάζομαι είσαι αρκετά δυνατός για να επιβιώσεις. Είναι επικίνδυνη αυτή η θέση εδώ δίπλα στην Περβάνσου. Να ελέγξουμε. Για την 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Voted. Yes, Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Για την 12 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 24 υπέρ, 23 κατά. Συμβαστική τροπολογία Β. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Δ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 έχει αποσυρθεί. 190 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 202 με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Να το ψηφίσουμε μαζί ή χωριστά. Μαζί. 202 συν την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.14, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42, υπέρ, κατά, αποχές. Α, τώρα πρέπει να ελέγξουμε για τη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. συμβασική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. συμβασική τροπολογία H υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 232 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία Ι. Α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία J. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 253 με προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ψηφίζουμε και για τα δύο μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία Κ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. όχι, τροπολογία 260 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 261 με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Ψηφίζουμε την 261 συν την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία L. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 268. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συγγνώμη. Σαΐντ. Ιδεολογικές σκέψεις. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Ε, για την 80 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 80, άρχεται η ψηφοφορία. πέρασε τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Οι 85 και 86 έχουν αποσυρθεί έχουν καλυφθεί. Συμβαστική τροπολογία M υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, α, καταπίπτει. 100 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά. Πάλι 103 υπέρ, κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Για την 103 άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Νόμιζα ότι είχε απορριφθεί. 105 υπέρ. Κατά αποχές ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασική τροπολογία όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασική τροπολογία π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την αιτιολογική σκέψη 12, 123 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία R υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 και 9 υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνονται. Είναι ταυτόσιμες. Για τις επόμενες μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. 70, 71, 72 και 73 on block. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία Εγκρίνεται 44 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και περνάμε στην ψηφοφορία για το τέλος των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Και αυτό είναι με ονομαστική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων, κατά, αποχές. Α, πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ναι, ναι, γι' αυτό έκανα και εγώ την ερώτηση. Αρχίζει η ψηφοφορία για την απόφαση να αρχίσουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 4 κατά. Ισχυρή εντολή λοιπόν προς την ομάδα που θα κάνει τις διαπραγματεύσεις. Και η τελευταία ελπίζω ψηφοφορία γιατί σε έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εισηγητής ο κύριος Κίρτσος. Ξεκινάμε με την συμβαστική τροπολογία Α. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασική τροπολογία C υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να το ελέγξουμε. Για την 84 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. πέρα της πληροφορία. Απορρίπτεται. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για την 1. Συμβαστική D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε. 105, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ίντα 18 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ψηφίζουμε για την 18 τη Ίντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έψηφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, δεν ήταν εύκολο να το δούμε, μικρή διαφορά. Συμβαστική τροπολογία H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο Budget. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Budget 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Y, Υπέρ. Α, έχουμε και μία προφορική τροπολογία. Αρχίζουμε με την ψήφιση της προφορικής τροπολογίας. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία και τη συμβαστική τροπολογία I, Ι, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αυτή είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία. Τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 1 με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 123 υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία για την 123. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά να το ελέγξουμε για την 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7 από μεταφορών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K β υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 2,60, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές. Πάλι δεν βλέπω καλά τη διαφορά. Ας ψηφίσουμε για την 2,60. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. Εγώ ρώτησα αν είχαν ψηφίσει όλοι, γιατί είδα ότι κάποιος μπορεί να μην... Ε, τώρα απερίφθη, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Οι κανόνες είναι σαφείς. 2.57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία ΚΒ2 με την προφορική τροπολογία. Ξεκινάμε με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία για την ΚΒ2. Εψήφισαν όλοι. Και η Σιλβία αυτή τη φορά. Θα σε φροντίζω, βλέπεις. Πέραση της ψηφοφοριες εγκρινεται εγκρίνεται. Τώρα, ΚΒ2 μαζί με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2.95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 302 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 306 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 3 και 4 δεν τις ψηφίζουμε. Είναι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές Ας ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 155. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έξι της ΔΕΒΕ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίγοι σοσιαλιστές παραπάνω για να καταλάβω κι εγώ καλύτερα τι γίνεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ. Ευχαριστώ, περβάς, Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία M υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ίντα 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία N υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ίντα 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ίντα 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία όμικρον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία π, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.18 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία R υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία TAF υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.34 υπέρ κατά αποχές. Να την ψηφίσουμε. 234. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο τη επικεφαλίδας 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιου. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 239. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 242 κατά αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ κατά αποχές απορριφθήκε 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριφθήκε 252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Την 252 ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφορίας. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 253 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 2.54 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίφθηκε. 255 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Πάντα η ίδια πλειοψηφία. Για να σας δώσω μια εικόνα. 2.56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα σιγά σιγά κουράζομαι. 262 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 263 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία όπως ελέγξαμε. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστευτείτε με τραν 3 υπέρ κατά. Εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Είναι τα 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D. Β μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 267. 267 γιατί γράφετε 268. 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, απορρίπτεται, συγγνώμη. Μπάτζεται 7 και 8 που δεν ψηφίσονται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. DV3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DV5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DV13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ιντα 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική χ υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 2,74 υπέρ. Περβάς, είσαστε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2,75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά. Είστε υπέρ. Ε? Ο Μπούρκαρτ είναι κατά. Πώς γίνεται. Ψηφίζουμε. 9-11 λοιπόν. Ψηφίζουμε. Και περάσαμε. 19-21 απορρίφθηκε. Την άλλη φορά να μου δώσετε λίγο παραπάνω ώρα. Ε, εγώ δεν πατάω κανένα κουμπί, δεν φταίω εγώ. Το είδα ότι απορρίφθηκε. Πολύ ωραία. ΔΕΜΠΕ 15 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Είναι τα ένα υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Είναι τα δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα τρία υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Είναι τα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 280 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ψηφίσουμε. Την 280 παρακαλώ ηλεκτρονικά ελέγχουμε. Πέρασε. Αν ψηφίσατε όλοι, απορρίφθηκε. Ευχαριστώ, μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω. Αρχικό κείμενο της Α, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Y, Y, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική Z, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 300... Α, συγγνώμη, συμβαστική Z, bis, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίφθηκε. Είναι το 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Είναι τα 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγράφος 30 αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις συντολογικές σκέψεις, συμβαστική ΑΑ. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο σε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική αβ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές απέχεται ή καταψήφισετε. Τότε θα χρειαστεί έλεγχος. Ηλεκτρονικός για την 25. Ψηφίζουμε. Έναρξη. Και αν ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίφθηκε και αυτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική ΑΣΥ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορριφθήκε. Συμβιβαστική αλφα-δι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι. Εγκρίθηκε. Και περνάμε στη συμβιβαστική ΑΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 48. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αν ψήφισετε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. 49 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Ε, έχετε κανένα πρόβλημα. Στα γαλλικά, όχι. Όλα μένουν καλώς. Α, το ελέγξαμε. Αρχικό κείμενο σε ό,τι αφορά την εκλογική σκέψη 2. Ευχαριστούμε, Άλφρεντ. Δίκιο είχες. IF, AF, στο H, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίθηκε ο συμβασμός μου, η 54 υπέρ, κατά αποχές, απορριφθήκε, 55 υπέρ, κατά αποχές, απορριφθήκε, τραν α υπέρ, κατά αποχές, εγκρίθηκε, τραν b υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τρανσί υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Citation 1 αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τελογική σκέψη 2 αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές 3. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ Κάτα. Αποχές. Χρειάζεται έλεγχος εδώ στην τρία Παρακαλώ, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τρία. Αν ψηφίσατε όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Η ισοψηφία, κάτι ήξερα που ζήτησα. Η ελληνική ψηφοφορία απορρίφεται. Αρχικό κείμενο εκτιμώντας 3 και 4 από κοινού υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Α, χρειάζεται έλεγχο. Πολύ λυπάμαι. Για την τροπολογία 4 παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Αν ψηφίσατε λοιπόν όλοι, λέει ο Πρόεδρος, πέρασε της ψηφοφορία. Ε, ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε να δώσουμε ένα δώρο, αλλά όχι με την υποστήριξη της ομάδα του Παύλου. Εκτιμώντα 6 και 7. Αρχικού κειμένου, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αρχικό κείμενο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Εκτιμώντα 9 και 10. Μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν. καταπίπτουν και πάμε στην 9. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε 10 υπέρ. Υπερβάνους και αυτή υπέρ. κατά αποχές εγκρίθηκε. Αρχική 11-12-13 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. Ναι, Η 11 υπέρ. Κατά. Α, τι ωραίο. Ας το ελέγξουμε. Η 11 παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι. πέρασε. Έγκρισε και Δεν ήταν σαφές. Τελευταία. Πραγματικά η τελευταία του Παμπλό, η 12 υπέρ. Παμπλό, θα είστε ευτυχισμένοι στην Ισπανία κατά αποχέ. εγκρινηθήκε. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο πώς και Ψηφίζουμε παρακαλώ ανέξι ψηφοφορίας. everyone voted? Αν ψήφισετε όλοι. Όχι. Λυπάμαι. Αυτά μένουν τελικά στα πρακτικά. Αν θέλετε λοιπόν να φανεί στο μέλλον ότι έχετε ψηφίσει, τώρα να ψηφίσετε. Πέρασε. Εγκρίθηκε 37 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και 2 οι αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Κίρτσο. Και να δώσω τώρα την Προεδρία στην συνάδελφό μου, προκειμένου να υπάρχει και gender balance στην Προεδρία, την Κέιτε και There's, there's been a terror attack. Υπήρξε μια τρομοκρατική επίθεση στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι με μεγάλη χαρά ως Προεδρεύουσα σήμερα για δεύτερη φορά θα καλωσορίσω την Έλκε Κιόνινγκ. Είναι εκπρόσωπος, πρόεδρος μάλλον του SRB, του Συμβουλίου Εξυγίανσης είναι η μόνη ομιλήτρια, οπότε θα έχει άνεση να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Είναι η πρώτη παρουσίαση της κυρίας Κέρνινγκ για το 17, ήταν μαζί μας το Δεκέμβριο του 2016. Σε επίπεδο SRB, Single Resolution Board, έχουν υπάρξει αποτελέσματα και βήματα προόδου και σε σχέση με το TILAP και σε σχέση με το MRL. Λοιπόν, με χαρά θα σας ακούσουμε, Πρόεδρε, γύρω στα 10 λεπτά και μετά να ζητήσω, παρακαλώ, ε, να σεβαστούν τα 5 λεπτά οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είμαι εδώ σήμερα, ένα χρόνο μετά αυτή την πολύ θλιβερή ημέρα για τις Βρυξέλλες και από ό,τι ακούω δυστυχώς θα είναι μια θλιβερή μέρα και για το Λονδίνο. Λοιπόν, ας περάσουμε στο πλαίσιο μας. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω το που βρισκόμαστε σε σχέση με την δημιουργία της υπηρεσίας μας και τα λοιπά, ε, Παντώ τις ερωτήσεις σας εκ των υστέρων αν θέλετε. Να πω ότι από την κρίση που ξεκίνησε εδώ και 10 χρόνια, το 2008, Πολλά έχουν αλλάξει, έχει ενισχυθεί η εποπτεία, έχει προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες μορφές, οι κεφαλαιοκές απαιτήσει έχουν ε, αυξηθεί, δημιουργήθηκε η Τραπεζική Ένωση και ένα νέο σύστημα εξυγίανσης ε, υιοθετήθηκε και συζητάμε ακριβώς ε, το καθεστώς αυτό των, της εξυγίανσης και ανάκαμψης και για τους κεντρικούς για τα CCP σε περιπτώσει. Έγινε μια μελέτη πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία λέγει ότι μεγάλες 26 ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να επιβιώσουν χωρίς επιμολύνσεις και φαινόμενα χιονοστιβάδας αν μία από αυτές αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που δείχνει ότι από την κρίση μέχρι σήμερα άλλαξαν τα πράγματα ε, και έχουν καταστήσει τα πιστοτικά μας ιδρύματα πιο ανθεκτικά και λιγότερο διασυνδεδεμένα. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ε, καταλαβαίνουμε ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα παλαιά προβλήματα σε ορισμένες χώρες ε, και πως η μετάβαση στο νέο πλαίσιο είναι μια δύσκολη μετάβαση για τις τράπεζες και τις αγορές κεφαλαίων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όμως τα θέματα αυτά να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν χωρίς το συνολικό πλαίσιο της ε, Τραπεζικής Ένωσης και να τεθεί ε, σε, κίνδυνο. Η κυρία Νουή θα σας μιλήσει αύριο για τα θέματα εποπτείας. Νομίζω πάντως ότι όχι μόνο είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την αποτυχία μιας τράπεζας, αλλά μπορούμε να πούμε με εμπιστοσύνη ότι οι περισσότερες τράπεζες στην Ευρώπη σήμερα είναι σε τέτοια κατάσταση που η αποτυχία τους δεν θα έφεται σε κίνδυνο την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και μπορούν να εξηγιανθούν εφόσον αποτύχουν όπως και άλλες ε, υπερχρεωμένες ε, εταιρείες στις υπόλοιπες αγορές. Ταυτόχρονα το επιπλέον δίκτυο ασφαλείας της εξυγίανσης που έχουμε στη διάθεσή μας είναι κάτι το οποίο είναι πράγματι διαθέσιμο ιδιαίτερα για τις αγορές οι οποίες επηρεάζουν τις αγορές. Θα χρησιμοποιηθεί το μέσο αυτό παρά μόνο, όταν είναι χρήσιμο για το ε, κοινό συμφέρον. Ε, και πρέπει να ασχοληθούμε τώρα και με θέματα που άπτονται περισσότερο βέβαια και του πτωχευτικού δικαίου, αλλά να δούμε τι γίνεται με το MRL, με τις ελάχιστες απαιτήσει, τα ελάχιστα προαπαιτούμενα. Οι τράπεζες που θα μπορούσαν λοιπόν ε, να ε, μπουν σε διαδικασίες εξυγίανσης προτείνεται το MRL που είναι ένα τμήμα των διαδικασιών εξυγίανσης, είναι ο βασικός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των τραπεζών. Το 2016 κάναμε σημαντικά βήματα για να βελτιώσουμε την βιωσιμότητα των πιστοτικών ιδρυμάτων, ξεκινώντας να παρέχουμε συμβουλές για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και αναπτύσσοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το MRL. Ε, το βασικό συμπέρασμα της δουλειάς του SRB για τα MRL το 2016 ε, και μετά από μια ανάλυση 70 τραπεζών μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωζώνη δείχνει να έχει κάποια θέματα αλλά τα θέματα αυτά αν και σημαντικά είναι διαχειρίσιμα. Ε, το ποσοστό αυτό δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό όπως το είχαν υπολογίσει οι εμπειρογνώμονες στο παρελθόν. Είχαμε μιλήσει για 110 δις στην έρευνα, ε, μιλάμε από 100 με 200 δις ανάλογα με το πώς μετράει κανείς. Αυτό το περίφημο, η τρομερό 8% το όριο το οποίο είχαμε θέσει σαν στόχο, ε, νομίζω ότι αποτελεί ένα θέμα για πολύ λίγες τράπεζες, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις η εφαρμογή της κατεξουσιοδότηση πράξης εισάγει υψηλότερες απαιτήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος ανησυχίας. Όπως έχω πει πολλές φορές, το MRL όχι κάτω από 8% του συνόλου της έκθεσης είναι κάτι το οποίο θα απαιτηθεί και για τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Τραπεζική Ένωση έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμες. Ε, επαρκής δυνατότητα απορρόφησης ζημιών, γιατί αυτό είναι το MRL, μεταθέτει το ερώτημα από το ποιος πληρώνει ε, στους μετόχους και τους πιστωτές. Τίθεται βέβαια και το θέμα των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του MRL, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν τους επόμενους μήνες. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άπαξ και είναι σαφές ότι το υπόλοιπο του 17 και το 18 θα χρειαστούμε για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Νομίζω όμως ότι έχουμε και άλλους τομείς ε, στους οποίους θα δουλέψουμε εκτός από τα MRL. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την λειτουργική συνέχιση των κρίσιμων υπηρεσιών μετά από την εξυγίανση. Οι ικανότητες των τραπεζών να βρουν ρευστότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Εδώ όμως χρειάζεται να συνεργαστούμε με την Κεντρική Τράπεζα όπως και η πρόσβαση στις υποδομές των χρηματοπιστωτικών μέσων, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις αγορές, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το 2017 ε, θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε λειτουργικές τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε σταδιακά είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετό καιρό και θα πρέπει να κρατήσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει νομίζω είναι η στρατηγική της εξυγίανσης. Υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στο απολαπλά σημείο εισόδου και το ενιαίο σημείο εισόδου το θέμα είναι αυτά τα προγράμματα να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης, να μην υπάρχει ένα μέγεθος για όλους και αυτό να εξαρτηθεί από το μέγεθος της τράπεζας, από το νομικό καθεστώς, από το πτωχευτικό δίκαιο και θα πρέπει ε, εδώ να εντάξουμε και τα MRL στο εσωτερικό των πιστοτικών ομήλων και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και στο εσωτερικό της Τραπεζικής Ένωσης αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η στρατηγική αυτή να καταστεί λειτουργική. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, καμία διάκριση εις βάρος κρατών μελών που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Τώρα για το Single Resolution Fund, το SRF, να πω ότι εμείς έχουμε ε, για το 2016 ε, ολοκληρώσει κάποιες διαδικασίες. Θα πρέπει και δεν είναι κάτι το θα έλεγα επίγον να δούμε ποια θα είναι η επενδυτική, ε, το επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο θα κινηθούμε και ταυτόχρονα το δίκτυο ασφαλείας το οποίο ολοκληρώσαμε στις αρχές του 2017. Έχουμε νομίζω συμφωνίες τώρα με όλες τις χώρες μέλη. Κάποια σχόλια επίσης για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα εφαρμογής του ΤΙΛΑΚ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Νομίζω ότι εμείς ε, θεωρούμε ότι οι προτάσεις είναι πολύ καλές, έχουμε και ανησυχίες και ερωτηματικά σε σχέση με τις προτάσεις αυτές. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ε, τον πρώτο πυλώνα, ένα δηλαδή ε, εθελοντικό αν θέλετε MRL, μόνο ε, για τις συστημικές τράπεζες και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και θα υποστηρίξω και εγώ αυτά τα οποία ζητάει η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις τράπεζες ε, για το αν θα δημιουργήσουμε εδώ μια διάκριση, ε, απότομη μάλιστα, ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες, κάτι το οποίο χρειάζεται και για όλες τις τράπεζες, όχι μόνο για τις μεγαλύτερες ή τις συστημικές. Και νομίζω επίσης ότι αυτό το οποίο έχει επίσης σημασία είναι οι αρχές εξυγίανσης να έχουν την απαιτούμενη ευελιξία έτσι ώστε τα MRL να έχουν το σωστό μέγεθος και σχήμα και σε επίπεδο διάρκειας χρονικής επίσης και οποιαδήποτε πρόταση μειώνει την ευελιξία για τις αρχές εξυγίανσης είναι κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει ανησυχίες. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μου να τελειώσω λέγοντας ότι πολλά μένει να γίνουν ακόμα γενικότερα στην, στις πιστοτικές δραστηριότητες. Το SRB πάντως είναι ε, προετοιμασμένο ή μάλλον θα είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει μια διαδικασία εξυγίανσης εάν είναι κάτι το απαραίτητο. Ευχαριστούμε πολύ. Λόγω στην κυρία μέρους του ΕΛΚΑ. Θα ήθελα να μιλήσω και για την υλοποίηση του TILAC, της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών. Η τελευταία έκθεση μιλά για τη μη τήρηση ε, των ε, περιθωρίων που αυτό μπορεί να οφείλεται όχι σε ε, έλλειψη κεφαλαίου, αλλά σε μη επιλέξιμες οφειλές. Και χορηγείται και μια περίοδος χάριτος πριν από την εφαρμογή των κυρώσεων. Υπάρχει επιλογή μεταξύ του να έχουμε μια διάταξη στην νομοθεσία και κάποιο βαθμό διακριτικής ευχέρεια, ευελιξία όπως είπατε κι εσείς. Και όταν βλέπουμε τις τροπολογίες ε, για το CRD, βλέπουμε ότι έχει δώσει περίοδο χάριτος έξι μηνών η Επιτροπή και από ό,τι κατάλαβα δεν σας ικανοποιεί και τόσο αυτή η προσέγγιση. Η ερώτησή μου προς εσάς λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη σας, τι θα αποτελούσε καλή λύση για να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία και να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση για διοικητικά θέματα. Δεν έχετε ακόμη υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας με την Επιτροπή. Θέλετε να σχολιάσετε. Υπάρχει ελπίδα να υπογραφεί. Και όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του SRB, εκκρεμούν ακόμη δύο πράξεις κατά εξουσιοδότηση στην Επιτροπή. Θέλετε να σχολιάσετε πώς βλέπετε τη διεκπαιρέωση αυτών των δύο, ας τα αποκαλέσουμε, διοικητικά θέματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όταν μίλησα για την ευελιξία, αυτό που εννοούσα περισσότερο ήταν ότι ο αριθμός του MRL πρέπει να είναι ε, κατά περίπτωση Δηλαδή θα πρέπει να λέμε το MRL του ΑΒΓ ανάλογα με την διαρθρωτική πολυπλοκότητα του ομίλου. Και όταν μιλάμε για την περίοδο χάριτος, όπως πολύ σωστά την ονομάσατε, συμφωνώ, δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτό το εξάμεινο που έχει τεθεί. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι εντάξει έξι μήνες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ε, είναι λάθος επιλογή και να μην υπάρχει αρκετό καταβληθέν κεφάλαιο διάσωσης και ίσως ε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποια λύση για να μην είναι αυτόματο το εξάμεινο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα διότι κανείς δεν μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να ξαναβρει κεφάλαιο, αλλά θα πρέπει να δούμε και την κατάσταση της κάθε τράπεζας. Για το μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση να υπάρξει μνημόνιο συνεργασίας και ε, ούτε φαντάζεστε πόσα ερωτήματα έχουν οι δικηγόροι για το ποιος κάνει τι. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τον οποίο δεν έχουμε ακόμη μνημόνιο συνεργασίας. Τέλος, για τις διοικητικές διαδικασίες, όντως είμαστε σε μια λεπτή θέση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει την κατεξουσιοδότηση πράξη για το πώς γίνεται η ανάκτηση των διοικητικών δαπανών του SRB από τον κλάδο. Μέχρι τώρα έχουμε ένα προσωρινό σύστημα και κατά βάση οι τράπεζες που ήταν στο SSM το 2014 προχρηματοδοτούν το διοικητικό προϋπολογισμό του SRB και το τελικό σύστημα θα το έχουμε ελπίζω του χρόνου. υπερβάμψη Περές εκ μέρου ε, των ε, Σοσιαλδημοκρατών. Κυρία Κιόνι, θα ήθελα ε, να επανέλθω στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στην πρόταση ε, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, γιατί αυτή η πρόταση επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο ε, ξέρουμε ότι υπάρχει όταν υπάρχει η βούληση ε, να παρέμβουμε στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή ο ασύμετρος κίνδυνος. Αλλά η δύναμη της αγοράς και η συνεννόηση μεταξύ φορέων, που είναι άλλοι δύο κίνδυνοι, δεν αντιμετωπίζονται από αυτή την πρόταση. θα μπορούσαμε να βασιστούμε στην εμπειρία της Βρετανικής Τράπεζας που στην περίπτωση της Northern Hawks με ένα μεικτό προϊόν, ε, τη δημοπράτηση, ε, έδωσε ένα τελικά θετικό απολογισμό για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα μπορούσατε λοιπόν εσείς να μελετήσετε μια τέτοια λύση. Τώρα θέλω να επανέλθω σε ένα γενικότερο πρόβλημα. Ποιος είναι υπεύθυνο σε όλη αυτή την αρχιτεκτονική δομή που έχουμε καθιδρύσει. Δεν φαίνεστε να είστε ιδιαίτερα θετικοί προς αυτή την πρόταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Βλέπουμε ότι αφενός με μακροοικονομικά, ό,τι ξεπερνάει το επίπεδο της δικής σας εντολής, ε, είναι κάτι ε, όπου η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θα ήθελε να προσπαθήσει να επιλύσει το θέμα του υπολείπου αυτών των εξυπηρετούμενων δανείων με μια κακή τράπεζα. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που έχουν μια μακροοικονομική εικόνα και πώς βλέπετε το διάλογο με αυτούς που έχουν μια πιο μακροοικονομική εικόνα για την ανάγκη απορρόφησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Και για την ερώτηση του πώς θα πρέπει να κοιτάξουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό αποτελεί μια ανησυχία όλο και πιο μεγάλη για τις ειδικές τράπεζες. Το ακούσαμε και σήμερα το πρωί για να σχολιάσουμε όμως την πρόταση για την EBA. Όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν ένα κληροδότημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ προσωπικά πολύ αμφιβάλλω κατά πόσον μια πρόταση η οποία τα βάζει όλα σε ένα ευρωπαϊκό σακούλι θα έχει ωφέλη. Γιατί προφανώς υπάρχει πρόφαση και όρεξη των επενδυτών για, τεχνητα... για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Αλλά αυτό είναι τεχνικό για την EBA, ε, για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Υπάρχουν πολλές συζητήσει τεχνικές. Μία εξ αυτών κατά πόσον θα πρέπει να κινηθούμε για μια οικονομική, προς μια οικονομική αξία. σε αντίθεση με πραγματικέ πωλήσει. Δεν νομίζω ότι θα καθαρίσει του συλλογισμού αυτό. Και από πιο τεχνική, τακτική μάλλον άποψη, σύμφωνο ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε κατά πάσα πιθανότητα υποστήριξη των μικρών τραπεζών για να προχωρήσουν. Αλλά όπως ακούσαμε, δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ένα σύστημα όπου το κράτος και τα δημόσια χρήματα χρησιμοποιούνται αλλά δεν μπορούμε να δούμε πώς θα βγουν οι δημόσιοι πόροι. Εδώ έχω επιφυλάξεις. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό σημείο είναι πραγματικά η ανάγκη διαφάνειας ε, στα χαρτοφυλάκια αυτά και να βρεθεί ένα πλαίσιο για να υποστηριχθούν κυρίως οι μικροί θεσμοί δεν μπορώ να σχολιάσω την Northern Rock γιατί πολύ, με πάσα ειλικρινή σας λέω ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες για τη συναλλαγή αυτή. Ποιο είναι υπεύθυνο τώρα. Νομίζω καταρχάς οι τράπεζες. Η τράπεζα επόπτης τώρα αναλαμβάνει δράσεις και έβαλε την πρόταση της ECB. Και επίσης πρόκειται και για ένα θέμα για όλους μας. Προφανώς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθορίσει το πλαίσιο για την αρχή εξυγίανσης. Μια τέτοια τράπεζα ή ένας διαχειριστής ε, περιουσιακών στοιχείων μπορεί να συμμετάσχει στην εξυγίανση, αλλά αυτό δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα. Ελπίζω να μην χρειαστεί η εξυγίανση. Ευχαριστούμε. Μικέλ Βέγκας από την ΚΟΕ. Όχι, Θα επανέλθουμε στο Μικέλ. Ο κύριος Ούρτασον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ακούσαμε με ικανοποίηση ότι εσείς εμένετε στο συγκεκριμένο θέμα με τα MRL, αλλά η χρήση του TILAC είναι εύκολο να κάνει κανείς τον υπολογισμό αν εφαρμόσουμε τα κριτήρια του 18% και του 6,75% των, της έκθεσης, τότε οδηγούμεθα σε κάτω του 8% αποτέλεσμα. Μήπως θα έπρεπε οι φιλοδοξίες για το τίλακ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι υψηλότερες. Η δεύτερη ερώτησή μου σχετικά με την προληπτική κάλυψη των απαιτήσεων θα πρέπει εσείς να προσπαθήσετε να δείτε ακριβώς τι σημαίνει η διαδικασία uh, soft, το λεγόμενο soft guidance και βλέπετε ότι ακριβώς αυτό το επίπεδο είναι κάτι το οποίο έχει άμεσες συνέπειες και γι' αυτό δεν ξέρω τι νόημα έχει να το, να το επιδιώξετε σε αυτή την φάση. Ε, σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορείτε να αγνοήσετε την παρέμβαση των ε, εποπτικών αρχών. Η μεταφορά του τίλαξ στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το 18% συν 6,75 μόχλευσης είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το τίλαξ σαν ένα ελάχιστο επίπεδο και ένα πλαίσιο MRL στα πλαίσια του πυλώνα 1 και πολλές φορές δεν οδηγεί στο 8% και υπάρχει και ο πυλώνας 2 όμως, κάτι το οποίο η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να αποφασίσει βασιζόμενη στην αξιολόγηση κινδύνου την οποία κάνει. Γι' αυτό είπα ότι απαιτείται ευελιξία έτσι ώστε ανάλογα με τη συστημική σημασία και την περιπλοκότητα να μπορούμε να πούμε ότι εδώ πρέπει να θέσουμε βάρος, να ρίξουμε βάρος στον πυλώνα 2. Όταν έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλες ε, πιστοτικές, ε, με μεγάλους πιστοτικούς οργανισμούς, θα πρέπει να είσαμε σε ε, θέση ε, την Δευτέρα να έχουμε διαθέσιμα κεφάλαια έτσι ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της αγοράς και σε πρώτη και σε δεύτερη φάση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να πούμε ότι ο πυλώνας 2 δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό. Τώρα, απαιτήσει και κατευθυντήριες γραμμές για τον πυλώνα 2. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει εύκολα με τις κατευθυντήριες γραμμές πυλώνα 2 εφόσον τον παρακολουθεί από κοντά. Και εφόσον δεν σέβεται το πιστοτικό ε, ίδρυμα τις κατευθυντήριες γραμμές πυλώνα 2, να τις κάνει απαιτήσει ε, εφαρμογής ε, πυλώνα 2. Κοιτάξτε, είναι ε, λειτουργικό το μέσο αυτό, απλά απαιτεί από κοντά παρακολούθηση. Βάλει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο φορές το κοινοβούλιο αυτό έχει περάσει ψηφίσματα σχετικά με την Τραπεζική Ένωση έτσι ώστε να υπάρξει αύξηση των αρμοδιοτήτων της ενιαίας εποπτικής αρχής όπως επίσης και το επίπεδο του προαπαιτούμενου κεφαλαίου. Βλέποντας ε, τους προϋπολογισμούς των τραπεζών στην Ευρώπη βλέπουμε ότι κάποιες τράπεζες ε, είχαν 80% έκθεση και σε νότιες χώρες βλέπουμε συστημικές, συστημικές τράπεζες οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια, δηλαδή σε τρίτο επίπεδο έκθεση χαμηλή και πολύ υψηλή εξάρτηση από την πίστοση, από τον τομέα των πιστοτικών. Τώρα για το πιστοτικό σύστημα είναι σωστό να υπογραμμίζεται ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένα συστημικό πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο γιατί περιλαμβάνει κάποια assets τα οποία είναι δύσκολα υπολογίσιμα. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω πώς το σύστημα ενιαίας εξυγίανσης μπορεί να αξιολογήσει τους κινδύνους αυτούς κατά τη διάρκεια της εξυγίανσης και σε ποιο βαθμό μπορείτε να προτείνετε προγράμματα εξυγίανσης υγιή και αποτελεσματικά ενώ δεν μπορείτε να υπολογίσετε ε, τα στοιχεία τα οποία έχει το συγκεκριμένο πιστοτικό ίδρυμα. Εμείς έχουμε μια περίπτωση στην Ιταλία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς για... είναι σαν να μην υπάρχει βούληση να δείξουμε ποιο είναι το πρόβλημα ε, ενώ πρόκειται για κάτι το οποίο είναι συστημικού επίπεδου ε, δεκάδες εκατομμύρια και φοβάμαι ότι ε, στην Ευρώπη νομίζω ότι έχει ξεσπάσει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, εμείς όμως ασχολούμαστε μόνο με το πιστοτικό κομμάτι. Τα προσιακά στοιχεία επίπεδο 3 αποτελούν ένα ζήτημα το οποίο οι επόπτες, δηλαδή το SSM στην προηγουμένη περίπτωση, παρακολουθούν πολύ στενά, είμαι βέβαιη και τον κίνδυνο πίστοση που συνδέεται και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι κατεξοχήν για τους επόπτες. Σημαντικό. Και για τους ε, λογιστές. Προκειμένου να είναι και να περιλαμβάνουν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όντω πρέπει να συγκαταλεχθούν στην κατηγορία 3, στο επίπεδο 3. Και από την προηγούμενη μου εμπειρία, σα το βεβαιώνω αυτό. Και έλεγχο έναντι των πραγματικών πωλήσεων και παρακολούθηση όταν βγουν από την κατηγορία αυτή τα προσιακά στοιχεία. Είναι σίγουρα αποπτικό ζήτημα, είμαι βέβαιη και συμφωνώ μαζί σα. Και προφανώ το πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν σχεδιάζουμε την εξυγένση. Ε, χρειαζόμαστε και τη διαφάνεια, χρειαζόμαστε και τα στοιχεία για του υπόπτε και για του οποίου θα πρέπει να δημιουργήσουμε δικλείδε ασφαλεία όπως και για τα χρωτοφυλάκια των MPL, ε, το μη εξυπηρετούμενο νέων. Για να δούμε δηλαδή προς τα ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται και το τι θα εφαρμοστεί σε περίπτωση εξυγίανσης. Δεν υπάρχουν θαύματα. Είναι και τα δύο προσιακά στοιχεία δύσκολα να αξιολογηθούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόκμαρκα. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη κύριε Χόκμαρκα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το χρόνο. Ο κύριος Βάλη θα κάνει μια ερώτηση. Έχω ένα λεπτό ακόμα, πρόεδρε, να κάνω την επερώτησή μου. Εξακολουθεί να είναι ασαφέ το πώ θα γίνει η εκτίμηση, γιατί επί τη αρχή αυτό που μπορεί να συμβεί είναι το εξή. Μπορεί να προκληθεί απόλυτη αξία των προϊόντων αυτών στην αγορά σημαντική, γιατί μιλάμε για όγκο πολύ ψηλότερο από τον ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων και μια και αυτό αφορά τα ιστορικά ε, μοντέλα των τραπεζών. Να ρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει άμεση επικέντρωση στα συστήματα αυτά, γιατί είναι πραγματικά κρίσιμη σημασία να επικεντρωθούμε σε αυτά. Και παράλληλα αυτά, όταν μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα, όταν μιλάμε μάλλον για σοβαρά προβλήματα, το οποίο είναι λιγότερο πρόβλημα από το, το, το, μη εξυπηρετούμενων δανείων, ε, επικεντρώνεστε και ανταποκρίνεστε πιο άμεσα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην απάντησή μου το διευκρίνησα αυτό. Θα το επιλύσει ο επόπτης. Γιατί ο επόπτης διαρκώς παρακολουθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία και σίγουρα δίνει έμφαση στα στοιχεία επίπεδου 3 ως θέμα ε, επικινδυνότητας της αγοράς και στα MPL γιατί συνδέονται με πιστώσεις. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε και μάλιστα με πολύ προσοχή. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και ζητώ συγγνώμη τον κύριο Χόκμαρκ που δεν είχε κοιτάξει την ώρα. Έχετε τώρα το λόγο. Δεν υπάρχει πρόβλημα να... Πρόεδρε, με την ευκαιρία αυτή κάνω και λίγο εξάσκηση. Όταν συζητήσατε το σχεδιασμό των τον MRL, είπατε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκές κεφάλαιο. Και προφανώς Αυτό ασφαλώ έχει να κάνει με το κεφάλαιο στην τράπεζα, το οποίο θα πρέπει να διτίθεται. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Ο επενδυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι διατρέχει κίνδυνο και από αυτήν την άποψη νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην υπάρχει οποιαδήποτε εικασία ότι υπάρχει κάποιο ποσοστό του κεφαλαίου το οποίο είναι διασώσιμο και κάποιο άλλο όχι. Και θα θέλω να επανέλθω στο σημείο αυτό. Και ε, να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κατάσταση προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η αυτόματη οίκαση, ότι κάποιο κεφάλαιο προορίζεται προς διάσταση και κάποιο άλλο όχι. Δεύτερη ερώτηση. Αν θα θέλετε να διευκρινίσετε κάποιες από τις ε, σκέψεις για το πώς έχει συσταθεί το BRD σήμερα η τράπεζα έρευνες και ανάπτυξης. Πείτε μας κάποιες σκέψεις σε ό,τι αφορά το Τίγλα και το MRL και την, ε, το ρόλο της BRD. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Μία από τις χειρότερες παρανοήσεις ήταν το γεγονός ότι ο κόσμος είχε την αίσθηση ότι κάποια στοιχεία θα ήταν υποδιάσωση. Και εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρώτα ήταν τα, η αρχή ήταν εξή, equity, junior bonds, μετά. Κανείς όμως δεν είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τις ε, senior bonds, τα ομόλογα αυτά. Το άκουσα αυτό πολλέ φορές, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτά. Και προφανώ. ότι τα τραπεζικά ομόλογα δεν έχουν να κάνουν με το ποιο είναι ο κάτοχο, έχει να κάνει με την κατηγορία στην ιεραρχία. Για να μην ρεαλιστέ όμω, αυτό που χρειάζεται και αυτό που περιλαμβάνεται στην πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα βήμα προ την κατεύθυνση είναι να διαπιστώσουμε ότι στην ίδια κατηγορία πιστωτών έχουμε και senior bonds, αλλά έχουμε και κάποιους πιστωτές, οι οποίοι για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να τους ε, διασώσουμε. Λειτουργική λοιπόν ευθύνη. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα πρέπει, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη και πιο διαφανής ιεράρχηση των πιστωτών, να υπάρχει μια τρίτη κατηγορία η οποία τώρα ενδεχομένως εξετάζεται. Κατά πόσον θα ιδρυθεί κατά πόσον θα ακολουθήσουμε κάποια άλλη ιδέα για να είναι σαφέ τι είδου ιεράρχηση θα ακολουθηθεί και αυτό θα πρέπει να το αποκαλύψουμε και να το δημοσιεύσουμε και στην αγορά για να το εκτιμήσει. Άλλα θέματα για την BRD. τίθεται ένας, ε, το θέμα του κανόνα ε, για την ε, υποταγή και το θέμα των, του ΤΙΛΑΚ. Τέλος, υπάρχει πιο πολύ ανάγκη όχι μόνο στην BRD, αλλά γενικά για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν με τα χάσματα που υπάρχουν στους εθνικούς νόμους, στην εθνική νομοθεσία για την αφαιρεγκαιότητα. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα θέξουμε και ενδεχομένω να δείξουμε την γενναιότητα, να δούμε εξειδικευμένου κανόνες αφαιρεγκαιότητα για για τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό κλάδο. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από τον Γιάκο Φονβάης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, Η πρώτη ερώτηση συνεχίζει um, την ερώτηση του Γκούνα που ρώτησε για τον Μπέιλιν. Um, Αν δούμε τι κάνουμε σήμερα στην Ευρώπη με τις μεγάλες τράπεζες, κάνουμε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση για να αποφύγουμε σοβαρές μορφές διάσωσης με ίδια μέσα και το κατανοώ αυτό. Συζητούμε την έννοια της δημιουργίας μιας κακής τράπεζας για να αποφύγουμε σοβαρές μορφές bail-in. Η ερώτησή μου είναι υπό ποιες συνθήκες νομίζετε ότι εξυγίανση με bail-in πιστωτών είναι προτιμότερη. Και πότε θα μπορούσε να είναι μετοχικό κεφάλαιο το εμπλεκόμενο στο bail-in. Άλλη μια ερώτηση, η εξυγίανση ενός σημείου εισόδου έναντι πολλαπλών σημείων εισόδου. Η ερώτησή μου είναι μήπως αν το κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, μήπως θα πρέπει να ξεχάσουμε την, ε, το ενιαίο σημείο επαφής ε, και να ε, έχουμε περισσότερες χώρες, κάτι το οποίο θα μπορούσατε εσείς να οργανώσετε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει προληπτικές κεφαλαιοποιήσεις. Είναι όμως ένα μέσο το οποίο έχει προϋποθέσεις και απαιτήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και νομίζω ότι είναι λογικό σαν μέσο σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχει κανείς την εντύπωση ότι όσο πιο κοντά έρχεται στα θέματα αυτά, λένε ότι το bail είναι ε, κάτι το οποίο βλάπτει την οικονομία και είναι φυσικά κάτι το βλαβερό, γιατί είναι σαφώς μια εξυγίανση, δεν είναι μια ανάσταση, κάποιοι χάνουν στοιχεία ιδιοκτησιακά. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό να, να αφορά το κεφάλαιο, αλλά και στα πλαίσια του πλαισίου α, κρατικής βοήθειας. Comment, ε, in saying τίθεται το θέμα του δευτερεύοντος χρέους και πράγματι αυτή η έκθεση είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποστεί ένα πρέπει να υποστεί το bail αλλά να δούμε και πού υπάρχουν παλαιού τύπου της προηγούμενης κατάστασης στοιχεία, κάτι το οποίο στα πλαίσια του φέντε θα χαρακτήριζε κανείς ακατάλληλοι επενδυτές. Έχουμε λοιπόν και εκεί κάποια θέματα. SPE για MPE εναντίον του e. MPE. Ενιαίο σημείο ή πολλαπλό σημείο εισόδου. Είναι θα έλεγα κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι λογικό στα πλαίσια της διαφάνειας. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές οντότητες στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και στο εσωτερικό της Ευρώπης και όλες είναι πάρα πολύ μικρές έτσι ώστε να τεθούν υπό τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Έχεις μια ποικιλία λοιπόν εποπτείας όπως και μια ποικιλία αρχών εξυγίανσης. Συνεπώς λοιπόν εδώ μπορεί να έχει κανείς ένα πιο διαφανή τρόπο εποπτείας, επίβλεψης και εξυγίανσης και εδώ νομίζω είμαστε σύμφωνοι με την αξιολόγηση που κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν αυτό είναι αντιθετικό με το SPE, ναι. Αλλά όπως είπα πριν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για 100% single point of entry και 100% MPE πολλαπλό ε, σημείο εισόδου. Συνεπώς λοιπόν ένα πολλαπλό SPE ή ένα MPE ενιαίο, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί σαν πιο ρεαλιστικό σενάριο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα πιστοτικ, ορισμένους πιστοτικούς ομίλους. Έχουμε επίσης κάποιες οντότητες εξυγίανσης οι οποίες ε, και αυτές δεν λειτουργούν με ενίο τρόπο, γι' αυτό καταλήγουμε πάντα σε μικτές μορφές αντιμετώπισης. Ευχαριστώ κυρία Κόνιχ και κυρία Ντελάγκε. Δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά το τίλακ. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τις ανησυχίες σας σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το κενό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στο ΤΙΣΕΠΣ e και τις υπόλοιπες τράπεζες, τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τύπων τραπεζών. Και εκφράσατε μια συγκεκριμένη ανησυχία, δεν ξέρω τι βάρος να δώσω. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για τα τύψιψ e ε, αντίστοιχο με τις ε, συστημικές τράπεζες ή κάτι ε, χαμηλότερων απαιτήσεων. Μία τράπεζα όπως η Monte και η dei η οποία δεν είναι συστημική, δεν θεωρείται, παρόλα αυτά θα μπορούσε να δημιουργήσει υψηλότατες πιώσεις, πιέσεις προς το πιστοτικό σύστημα στο σύνολό του. Και για το ίντες επίσης, ξέρετε ότι ε, και εμείς η, η ομάδα των σκιωδών το συζητάμε το θέμα, υπάρχει πρόοδος και μιλάμε για χώρες όπου το επίπεδο προστασίας δεν είναι αντίστοιχο με αυτό το οποίο προβλέπει το AIDS. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι κάποια πιστοτικά ιδρύματα από τρίτες χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται με τις εθνικές EDS, GDS εφόσον δεν είναι αντίστοιχο το επίπεδο προστασίας στη χώρα προέλευση. Συμφωνείτε με την αντίληψη αυτή. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σας βοηθήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να ελέγξουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τις ισορροπίες οι οποίες υπάρχουν. Θα ήθελα μια πρώτη αντίδραση τώρα και θα ήθελα για το θέμα αυτό να μείνω σε επαφή μαζί σας αργότερα. Ξεκινώντας με την πρώτη παρατήρηση, πιστεύω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε για το TILEC το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των G-SIPs. Αλλά θα πρέπει να δούμε σε όλες τις χώρες ότι η, στρατη... συστημική σημασία και οι... Οι... οι τράπεζες οι οποίες είναι ε, μικρότερη σημασίας, στη δική μου ας πούμε η Commerzbank και η Deutsche Bank είναι συστημικές. Ανησυχούμε όμως ότι ε, με τον πυλώνα ένα μόνο για τις τράπεζες αυτές είναι πολύ σκληρός ο αγώνας έτσι ώστε να καταλήξουμε στο ίδιο MRL και με τον πυλώνα 2. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν προτιμότερο να πούμε ότι αυτό αφορά μόνο τις ε, εσωτερικά σημαντικές ε, τράπεζες ή μήπως να πούμε ότι μιας και δεν υπάρχει για αυτές τις τράπεζες πυλώνας ένας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες απαιτήσει MRL. Στην ουσία δηλαδή το θέμα παρουσιάζεται με μεικτό τρόπο και εγώ θα ήμουν πάντα υπέρ της υποχρεωτικής, του υποχρεωτικού πυλώνα 1 για τις συστημικές τράπεζες, για το ίντες. Εγώ βλέπω ποια είναι η ανησυχία σας και πράγματι Υπάρχει και ανησυχία στο εσωτερικό της ε, Τραπεζικής Ένωσης και της Ευρώπης. Βλέπουμε ας πούμε ορισμένες περιπτώσεις όπου ε, κάποιες, ε, κάποιες τράπεζες ανοίγουν παραρτήματα σε άλλες χώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πίεση θα έλεγα και στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων της χώρας προέλευσης αν θέλετε της τράπεζας και αυτό ε, πολλές φορές, αυτή πολλές φορές είναι η μικρότερη χώρα ή η ασθενέστερη χώρα ή λιγότερο ισχυρή εν πάση περιπτώσει χώρα σε επίπεδο προστασίας καταθέσεων. Ε, μπορεί να διαρωτηθεί κανείς αν γνωρίζουν ακριβώς τις ε, δραστηριότητες του τραπεζικού αυτού οργανισμού σε άλλες χώρες. Είναι δύσκολο λοιπόν να φροντίσει κανείς το θέμα αυτό και να αναζητήσει τις αντιστοιχίες. Είναι κάτι, ε, όταν μιλάω για αντιστοιχίες ξέρω τι σημαίνει και ξέρω τι προβλήματα δημιουργούνται και γι' αυτό η πρότασή σας να το ξανασκεφτώ μου ταιριάζει. Ευχαριστώ. Τέλειωσα τον κατάλογο των ομιλητών. Σε μια διαδικασία κατστιάει τώρα. Υπερβάζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα θέλω να επανέλθω σε κάτι που είπατε σήμερα το πρωί. Είπατε ότι ε, μιλήσατε για μια περίπτωση διαμεσολάβησης. Υπό ποιου όρου λοιπόν ο μηχανισμός αυτός, ε, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί ω τώρα, κατ' εξαίρεση ουσιαστικά, πώς λειτουργεί λοιπόν και υπό ποιου όρου, Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση λοιπόν. Ήταν ε, δύσκολη φαντάζομαι η πλειοψηφία στο σώμα και ποιε ε, ήταν τα συμπεράσματα που εξαγάγατε προκειμένου να μπορεί να κινητοποιηθεί πιο εύκολα ο μηχανισμό αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Η Εστέντε ναι, Λάγκε αναφέρθηκε στο ΕΝΤΙΣ και οι συζητήσει στο Συμβούλιο ξεκίνησαν σε ό,τι αφορά backstop. Έχετε επιπρόσθετα στοιχεία να μας παρουσιάσετε για την εξέλιξη του μωρού αυτού. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω από τα θέματα διαμεσολάβησης. Οι όροι για να ξεκινήσει αυτή η διαμεσολάβηση και το ξέχασα αυτό στο πλαίσιο του ΕΣΜΑ, είναι λίγο διαφορετικές σε περίπτωση σωμάτων εξυγίανσης, αν μία από τις αρχές δεν είναι ικανοποιημένη με το σχέδιο εξυγίανσης και θεωρεί ότι υπάρχει ένα σημείο όπου δεν αποτυπώνεται κάτι επαρκώς. Μπορούν να καλέσουν την EBA για διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο εμπόδιο και δεν χρειάζεται υπερβολική, μάλλον ειδική πλειοψηφία για να περάσουμε σε διαμεσολάβηση. Τον έφερα σήμερα το πρωί για δύο λόγου. Κοιτώντα όλα τα μέσα τα οποία έχουν ε, συμφέρον στο CCP, στην ανάκαψή και στην εξυγίανση ή εν πάση περιπτώσει στην περίπτωσή μου για την εξυγίανση, θεωρώ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε σχέση με τα σώμα. Όλοι θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και θα πρέπει να συμφωνούν. Και αν δεν συμφωνούν θα πρέπει να υπάρξει διαμεσολάβηση. Άρα το εμπόδιο θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από αυτό που ανέφερε στο τύπημα Γιώργη σήμερα το πρωί. Για το άλλο ζήτημα Νομίζω ότι θα συμφωνούσε κατά πάσα πιθανότητα η Esther Delange ότι το ΕΔΙΣ κινείται αργά. Αργά αλλά κινείται. Και για τον backstop να πω ότι μόλις ξεκίνησε να μετακινείται. Στο Συμβούλιο αποτελεί θέμα εργασίας, κοιτάνε τις τεχνικούς όρους ενός backstop, αλλά σίγουρα θα πάρει χρόνο. Και εμείς πάντα λέγαμε ότι Εργαστήκαμε σκληρά για να υπάρξουν συμφωνίε διευκόλυνση των δανείων, αλλά προφανώ θα πρέπει να υπάρχει αυτό το backstop και συμμετέχουμε λοιπόν στην εργασία αυτή. Δεν φαντάζομαι βέβαια να το ολοκληρώσει η Μαλτέζικη Προεδρία. Και ούτε καν και η Εστονική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, α είμαστε και λίγο αισιοδόξοι, δεν βλάπτει. Περιβάλλον, αν θέλει να κάνει επερώτηση. Θα ήθελα να μας πείτε για τις δικές σας εμπειρίες για τη διαμεσολάβηση. Υπάρχει το θέμα της εκκίνησης και το υπάρχει και το θέμα του πώς λειτουργήσε στην πράξη. Τι πληροφορίες έχετε εσείς και ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία εξάγαγετε. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς το βιώσατε. Νομίζω στη δική μας περίπτωση υπήρξε μια μεσολάβηση στην EBA και το θέμα ήταν ότι ένα από τα κρατημέλη είχε μεγάλες ανησυχίες για την προστασία μιας θηγατρικής στο κράτος και ότι οι ανησυχίες δεν αποτυπώθηκαν επαρκώς. Αυτό που μάθαμε είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα και ότι δεν μπορούμε απαραίτητα να προχωρήσουμε είναι λίγο μια διαδικασία in and out. Κατά πόσον τα ζητήματα αυτά είναι τόσο σημαντικά εσωτερικά τη Emerald. Κατά πόσον είναι λειτουργικά και κατά πόσον αυτό που υπάρχει στη θεωρία όντως λειτουργεί στην πράξη. Αυτό θα ήταν το βασικό θέμα. Η βασική μου εμπειρία δεν θα ήθελα πιστεύω να, μπω σε λεπτομέρειε. Μάλιστα, ολοκλήρωσαν τον κατάλογο αυτή τη φορά. Κάτσε τη αν θέλει κανεί το λόγο, ο Σβεν äh, Γκίγκολτ. ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κυρία Κιόνιχ. Θα μιλήσω αγγλικά γιατί είναι οι περισσότεροι αγγλόφωνοι από τους παρόντες. Έχω μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι σχετική. Γίνεται μια ευρεία συζήτηση και αντικατοπτρίζεται και στην αγορά ότι πολλές τράπεζες που η αγορά τις θεωρεί προβληματικές ή πιθανώς προβληματικές είναι τράπεζες που μπορεί να επιβλέπονται από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και πολλοί πολίτες έχουν αμφιβολίες για το αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεπερνάει τα όρια των ρυθμιστικών διατάξεων γιατί δεν δηλώνει ότι κάποιες τράπεζες που έχουν μεγάλο πρόβλημα μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν, δηλών δεν τις δηλώνει ως προβληματικές ή σχεδόν προβληματικές. Σας δώσαμε τώρα την εξουσία να αρχίζετε εσείς αυτή την ε, διαδικασία και το κάναμε επειδή ήδη είχαμε Πολλέ κακές εμπειρίε στο παρελθόν. Θέλω λοιπόν να σα θέσω το ερώτημα, εάν εξετάσατε ήδη σοβαρά κάποιες τράπεζες στο πλαίσιο της άμεσης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θεωρείτε ότι είναι πιθανόν, εάν σκέφτεστε το ενδεχόμενο, να ξεκινήσετε εσείς την διαδικασία εξυγίανσης. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι συζητήσατε στο SRB και πόσο έχετε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να δηλώσετε ε, ως προβληματικές τράπεζες κάποιες τράπεζες που έχουν μεγάλο πρόβλημα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναρωτιόμουν ποιος θα μου κάνει αυτή την ερώτηση και πόσο θα αργήσει. Σαφώς υπάρχει μια διπλή διαδικασία ενάψηματος ε, απαρχής της διαδικασίας και εξετάζουμε όλες τις τράπεζες και αυτές τις τράπεζες που βρίσκονται σε πιο επισφαλή ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έχει μια κατηγοριοποίηση και εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τον κατάλογο. Μέχρι τώρα νομίζω ότι είμαστε σε θέση όπου εμείς πρέπει να συμπεράνουμε ότι κάποιες τράπεζες έχουν ακόμη κάποιες ευκαιρίες και δεν είναι ακόμη προβληματικές. Η ανάλυση συνεχίζεται και θα είναι μια διαρκής ανάλυση, αλλά κυρίως οι επόπτες πρέπει να το κάνουν αυτό, γιατί οι επόπτες έχουν πιο ενεργές πληροφορίες. Εμείς ερχόμαστε δεύτεροι. Το εξετάζουμε, εξετάζουμε τις τράπεζες και αν ε, χρειαστεί θα δώσουμε το σήμα ότι πρόκειται για προβληματική ή πιθανώς προβληματική τράπεζα. Ο κύριος Γκίγκολτ. Έχετε ήδη εξετάσει λεπτομερώς μία ή περισσότερες τράπεζες και έχετε ήδη ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για να εξετάσετε ε, εάν οι αποφάσεις ή η μη λήψη αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ορθή κατά τη γνώμη σας. Δεν κάνω σχόλια σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σαφώς ε, παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή αρκετές ε, περιπτώσεις. Ο κύριος Γκίγκολ και πάλι. Μπορείτε να μας πείτε πόσες υποθέσεις εξετάζετε σε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Όχι, διότι όπως σας είπα είναι αρκετές υποθέσεις, όχι μία ή δύο. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Κένιχ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για άλλες ερωτήσεις και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση θα ήθελα να καταγράψουμε στα πρακτικά την ε, θλίψη μας για τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο σήμερα το απόγευμα. Τουλάχιστον δύο θύματα και αρκετοί ε, σοβαρά τραυματισμένοι χάρη στις υπηρεσίες, άμεση υπηρεσίες άμεσης επέμβασης ε, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και ένας από τους σοβαρά τραυματισμένους ε, είναι ένας ε, αστυνομικός εν υπηρεσία. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί στις 9 με την ετήσια έκθεση για τον ενίο υποπτικό μηχανισμό. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν.